Σα Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία και καθίστε. Να ξεκινήσουμε με την απογευματινή μας συνεδρίαση. Bueno. Pues a todos por... Καταρχάς σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την απογευματινή συνεδρίαση με τους υπόλοιπους προσκεκλισμένους μας για την ακρόαση για την Πράσινη Βίβλο για την ε, κοινή πολιτική αλίας. Θα αρχίσω να δίνω το λόγο σε όλους σας. Σας ε, παρακαλώ για άλλη μια φορά να τηρείτε τα χρονοδιαγράμματα. Καταρχάς έχουμε τον κύριο Armstrong, Διευθυντή τη Scottish Fisherman Federation που έχει το λόγο για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσει τη δική του άποψη για την Πράσινη Βίβλο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα περάσω κατευθείαν στη δήλωση όσον αφορά ως Ένωση Σκότων Αλλιέων. Ε, Φυσικά δεσμόβεσαι με τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΛΠ με τη σημερινή της μορφή την αξιοποίηση όλων των θελάσσιων πόρων μέσα σε βιώσιμα πλαίσια και το διαψάστη ομοφωνία το πρωί. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε όμως η συγκεντρωτική μικροδιαχείριση. Τώρα για την πράσινη, για την πράσινη βιβλία είναι απογοητευτικό το ότι δεν λαμβάνει υπόψη θετική δράση όπως είπε ο Σνάφος Παστόρ το πρωί ότι η πράσινη βίβλος υπάρχουν καλά παραδείγματα σχετικά με τη συμμόρφωση και με την καινοτομία όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τα οποία θα πρέπει, διατηρησιμότητα μάλλον, τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε κι άλλο, σχετικά με τον υπερβάλλοντο στόλο. Κατά την άποψή μας, τα μέτρα θα πρέπει να αφορούν μόνο περιπτώσεις όπου επηρεάζεται το απόθεμα θέματα οικονομικής ευελιξίας ή κοινωνικής βιωσιμότητας. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν ο πελαγικός στόλος της Σκοτίας που δεν εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις ποσοστάσεις της αλλά φροντίζει να κρατάει ακέραιο το, τις επιδόσεις όσον αφορά την διατηρησιμότητα. Τώρα, τα αλλιευτικά δικαιώματα και σχέση, σε σχέση με την υπεραλίευση. Τα διεθνώς εμπορεύσιμα δικαιώματα θεωρούμε ότι θα ήταν σε βάρος της ε, σκοτσέζικης, ε, του κλάδου της σκοτσέζικης αλλιάσης. η ΚΑΛΠ θα πρέπει να προβλέπει μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των αποθεμάτων και οικονομική βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις. Θέματα κοινωνικής διατηρησιμότητας καλύτερα να μείνουν στο καλύτερο επίπεδο διαχείρισης που είναι το εθνικό. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων δεν είναι ρεαλιστικό. και δεν ε, συμβαδίζει με τα επιστημονικά δεδομένα. Πρόκειται για ένα απλώς άθροισμα μέτρων. Αυτό δεν θα έπρεπε να παραμείνει στην αναθεωρημένη κάλπ. Τότε η μη συμμόρφωση και η ανευθυνότητα είναι συστημικά χαρακτηριστικά της αλλίας, δεν βοηθάει. Θα σας πω γι' αυτό λίγο μετά. Τώρα το πλαίσιο λήψης των αποφάσεων για βασικές αρχές. Θεωρούμε ότι η αποκέντρωση της διαχείρισης της αλλίας στο επίπεδο όσο πιο κοντά γίνεται στον συγκεκριμένο φορέα θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό του νέου μοντέλου. Διότι σήμερα με συγκεντρωτική γύψη των αποφάσεων αυτό είναι η πιο μεγάλη αποτυχία της ΚΑΛΠ. Το είπε ο Ιαν Μαξουίν το πρωί ότι μεταναστευτικά είδη που καλύπτονται από τα πελογικά ρακ και αλληστεύονται από τις πελαγικές αλλιευτικές μονάδες δεν ταιριάζουν με το αποκεντρωμένο μοντέλο. Συνεπώς δεν υπάρχει μία λύση για όλους όσον αφορά την αποκέντρωση. η ενθάρρυνση του κλάδου να αναλάβει περισσότερες ευθύνες στην εφαρμογή της διαχείρισης και της αναφερεμένης κάλπ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η εμπειρία επιβεβαιώνει ότι η ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον κλάδο διευκολύνεται αν παίρνει μέρος στις αποφάσεις. Σε συνεργασία με κίνητρα για να υπάρξουν μέτρα, γιατί αυτό είναι το σωστό, να γίνεται το σωστό. Αν επιβληθούν μέτρα θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και θα κάνει ζημιά στην ικανότητα του κλάδου να αναλάβει τις ευθύνες του. Ρυθμίζοντας τα του κλάδου φυσικά εμπεριέχει ένα στοιχείο κόστους. Και το να δημιουργηθούν κατάλληλες ε, κατάλληλοι οργανισμοί. Αυτό φυσικά θα σημαίνει κόστος στον κλάδο, αλλά είναι διατεθειμένος να το πληρώσει προκειμένου να παίρνει μέρος στη διαχείριση στο σωστό επίπεδο. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συμμόρφωσης. Και αυτό ισχύει με έναν κανονισμό ο οποίος να έχει συνέπεια και εφαρμογή του στο σωστό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αμείβονται αν πετυχαίνουν τους στόχους της και να υφίστανται κυρώσεις αν δεν το κάνουν. Τώρα, σε σχέση πάλι με κάτι που υπόθηκε το πρωί, διαφοροποιημένα αλλιευτικά καθεστώτα για να προστατεύονται οι μικροί παράκτη αλλιευτικοί στόλοι. Ξέρουμε και το ξέρουμε και στη Σκοτία, ότι η συγκεκριμένη συμβολή αυτό το μικρό στόλο που δεν είναι καθόλου μικρή η αναλογία του όγκου των ψαριών οι ευκαιρίες αλίευσης που έχουν και ο έλεγχος αυτών των μονάδων ποικίλει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Επομένως, θεωρούμε ότι η διαχείριση αυτών των στόλων είναι θέμα κράτους μέλους. Δεν μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά. Με μία λύση για όλους, την ίδια. Από τα μικρά σκάφη των διοικητικών αχθών της Σκοτίας μέχρι τους μεσογειακούς στόλους. Επειδή θέλουμε να αξιοποιήσουμε την αλληλεία. λέμε ότι αδιαμφισβήτητα οι ποσοστώσεις επιμέρους ειδών, προκειμένου να ρυθμιστεί μέσω αυτών μία αλληλεία πολλών ειδών, εμπεριέχει ε, αρνητικά στοιχεία. Ορισμένα τάξη και όλα αυτά τα ψάρια ψαρεύονται στο ίδιο δίχτυ. Μετά αν θέλουμε να τηρούνται οι κανόνες σύνθεσης και οι κανόνες του τάξη, σημαίνει κατά ανάγκη θα υπάρξει απόρριψη. Το είπαν αυτό οι ομιλητέ. Πρέπει στη μεταρρυθμισμένη κάλπ να βρούμε μια μέθοδο για την αλληλεία πολλαπλών ειδών με μεικτά αλλιεύματα. Η αλληλεία πολλαπλών ειδών και τα σχέδια ίσως είναι ένα πρώτο βήμα στη βελτίωση της διαχείρισης και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κλάδο να κάνει ορισμένα πειράματα για καλύτερη χρήση στην αλληλεία πολλαπλών ειδών. Δύο λόγια για το MSY. Η αρχή του MSY κακώς υπερεκτιμάται δεν ταιριάζει μια προσέγγιση οικοσυστημική, δεν είναι καλά ορισμένη, επειδή συμφωνήθηκε αυτή η αρχή σε πολιτικό όργανο, στο WSSD το 2002, υπάρχει υποχρέωση από τη στιγμή που υπεγράφει αυτό, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος ότι πραγματικά δουλεύει ως αλλιευτικό εργαλείο. Συμφωνήθηκε σε ένα πολιτικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν θέλουμε μια οικοσυστημική προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και άλλες θεωρητικές υποθέσεις όπως maximum οικονομική απόδοση ή η μέγιστη κοινωνική απόδοση και τα RACS θα μπορούσαν ενδεχομένω να φροντίσουν αυτές οι διαστάσεις να μπουν στα μακροπρόθεσμα προγράμματά τους. Το τελευταίο μείζον θέμα, δύο θέματα μάλλον, είναι η σχετική σταθερότητα η σχετική σταθερότητα είναι σημαντική με τη σημερινή της μορφή. Έτσι το θεωρούν οι Σκοτσέζοι Αλλιείς. Μπορεί να πει κανείς ότι εκπροσωπεί τα ιστορικά δικαιώματα πρόσβασης των κρατών μελών σε φυσικούς πόρους στα υδατά τους. Αν αλλάξουμε την σχετική σταθερότητα επηρεάζεται από αλλιευτικές ευκαιρίες του παρελθόντος. Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν και μπορεί να ανταμείβουμε κακή συμπεριφορά κρατών που δεν ρύθμισαν το στόλο τους σχετικά με την ικανότητά του να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έχει η χώρα. Και στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα θα αναφέρω την πολιτική που χαράζεται με βάση τις γνώσεις. Αυτό το συμφώνησε φυσικά η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία μας ότι είναι θεμελιώδης ενδιαφέρει όλους τους φορείς και θέλουμε να είναι μέρος των νέων προγραμμάτων. Κρατήθηκα στην ώρα μου, ευχαριστώ. 15 δευτερόλεπτα υπερβικά το χρόνο σα αν δεν πειράζει σας χώρα λέει η πρόεδρος. Είμαι αυστηρή, αλλά όχι και τόσο. Αυστηρή. Δίνω το λόγο στην κυρία Ούτα Μπελιών, που είναι η συντονίστρια του συνόλου της ε, ομάδας μάλλον των μη κυβερνητικών οργανώσεων όσοι 2012 για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είμαστε εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Είμαι η Διευθύντρια του Προγράμματος για τα Θαλάσσια Θέματα και είμαι συντονίστρια του Ocean 2012 που είναι μια ευρία, ένας ευρύς συνασπισμός μη κυβερνητικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται για τα θαλάσσια θέματα και για την προστασία των ωκεανών και εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στην μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Μια πλήρεστερη μορφή της παρουσίασής μου είναι διαθέσιμη στην είσοδο αυτή τη αίθουσα και στην ιστοσελίδα μα θα βρείτε ακόμα περισσότερα στοιχεία αν θέλετε να έχετε περισσότερε λεπτομέρειε, γιατί είναι λίγο ο χρόνο και θα εστιάσω μονάχα σε μερικά κομβικά σημεία. Οι πολίτε όλη τη Ευρώπη ενδιαφέρονται σε, για ένα σύνολο θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλία και τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Του ενδιαφέρει φυσικά η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντο που είναι κοινό κληροδότημα σε όλου μα. Του ενδιαφέρουν τα θέματα ανάπτυξη και τα κοινωνικά θέματα, θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία των παρακτήων κοινοτήτων, θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των προϊόντων που έρχονται στην αγορά και φυσικά τους ενδιαφέρει και η διαχείριση του χρήματος των φορολογουμένων και οι δημόσιες ενέργειες υποστήριξης προς την αλία. Όλα αυτά τα συμφέροντα λοιπόν έχουν συνασπιστεί σε ένα ευρύ συνασπισμό <clears throat> φορέων που απαρτίσουν την Ocean 2012 και έχουν σαν στόχο να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση μετά από το γεύμα κανείς ε, χαλαρώνει λιγάκι, αλλά εγώ προσπαθώ και πάλι να εστιάσω την προσοχή σας στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι λοιπόν, αυτό είναι το όραμά μας, θέλουμε να είναι υγιής οι ωκεανοί με πολλά ψάρια και ε, φυσική ζωή που συμβάλλουν στην ανθρώπινη ευμάρεια. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να επιτύχουμε αυτές τις αλλαγές που είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί το, αρκετά το γεγονός ότι η τωρινή κατάσταση δεν είναι παραδεκτή, ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση η οποία έχει ήδη διατυπωθεί από τον Επίτροπο κύριο Μπόρτς. Ελπίζουμε ότι και η κυρία Ταμανάκη όταν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει και αυτή, αυτή την ε, πρόκληση και θα προωθήσει ενεργά την αλλαγή προς μια βιώσιμη μορφή αλίας. Οι κύριες προτάσεις μας λοιπόν για μεταρρύθμιση ποιες είναι. Και θέλω να τις συνδέσω με το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δείτε αν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα υποστηρίζετε. Εμείς υποστηρίζουμε σαφώς να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα του περιβάλλοντος, στην επίτευξη στόχων του περιβάλλοντος. Γιατί είναι σαφές ότι χωρίς ψάρια δεν υπάρχει ψάρεμα. Αν θέλουμε να έχουμε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα <clears throat> και αηφορία θα πρέπει να θέσουμε σε πρωταρχικό επίπεδο την υγεία των αλλιευμάτων και των ωκεανών. Δεύτερο και εδώ ίσως μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά με την ε, έκθεση γιατί δίνουμε διαφορετική στοχοθεσία σε σχέση με τα θέματα αυτά. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ του στρατηγικού επίπεδου, του πολιτικού επίπεδου και του διαχειριστικού επίπεδου. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια για την αλίευση που να βασίζονται σε, επιστημονικές, σε επιστημονικά δεδομένα. Τα επιστημονικά δεδομένα όμως έχουν μια αξία που εξαρτάται από το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκπονούνται. Με ποια πιθανότητα λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την υγεία των ωκεανών μας. Ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Μας έχει κανείς ρωτήσει αν θέλουμε 88% των αλλιευμάτων μας να την χάνουν υπερεκμετάλλευσης και 30% από αυτά να είναι πέραν των βιολογικών ορίων. Δεν ξέρω αν ρώτησε κανείς τους πολίτες της Ευρώπης αν είναι αυτό αποδεκτό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σε επίπεδο Συμβουλίου και από σήμερα πια και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποια μακροχρόνια προοπτική, μια μακρόπνοα προοπτική σε σχέση με το ποιο πρέπει να είναι το στρατηγικό πλαίσιο της αλίας. Μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορούν να μας δώσουν τις συμβουλές τους οι επιστήμονες και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές τις συμβουλές. <clears throat> και εμείς δεν υποστηρίζουμε το να περάσουμε από τα όρια αλλιευμάτων στον περιορισμό της αλλιευτικής ικανότητας και μπορούμε να σας δώσουμε τα επιχειρήματά μας εγγράφως με πιο πολύ λεπτομέρεια και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σαφές και στη διαδικασία, μέσα στη διαδικασία διαβούλευσης επίσης. Θέλουμε ότι πρέπει να υπάρξει σαφή μείωση τη αλληλευτική ικανότητα. υπάρχει υπερβολική ικανότητα, Κανεί δεν ξέρει πόσο, σε ποιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει όμω ότι πρέπει να έχουμε και καλύτερη συλλογή στοιχείων και για μας είναι σημαντικό η μείωση της ικανότητας να μην είναι μονάχα ποσοτική αλλά και ποιοτική. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να γίνει πιο διάφανη και συμμετοχική. Και εδώ συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Αλλά θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει και να είναι κομμάτι των εμπλεκομένων και κάτι το οποίο ίσω είναι καινούριο σε αυτή τη συζήτηση, θεωρούμε ότι οι κανόνε πρόσβαση στα αλλιεύματα θα πρέπει να βασίζονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, εάν θέλουμε πράγματι να προχωρήσουμε προς καλή ποιότητα του περιβάλλοντο και βιώσιμη αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό το οποίο λέω. Τα κριτήρια τα οποία εμεί υποστηρίζουμε ιδιαίτερα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την επιλεκτικότητα. Αυτές οι μορφές λοιπόν ε, που οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο παραλιευμάτων θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητες. Αυτές που βλάπτουν περισσότερο το περιβάλλον θα πρέπει να ευνοηθούν. Πολλές φορές η αλία οδηγεί σε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι πολύ καλό σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, πραγματικά την κλιματική αλλαγή, για τις συνθήκες απασχόλησης και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για μας, μας ενδιαφέρουν τα κοινωνικά στοιχεία, μας ενδιαφέρει η ποιότητα του τελικού προϊόντος και φυσικά μας ενδιαφέρει και το ιστορικό της ε, συμμόρφωσης για όλα αυτά τα κριτήρια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς οι οποίοι εκπληρούν όλα αυτά τα κριτήρια στο μεγαλύτερο βαθμό και αυτό σημαίνει ότι θα μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους προς μια βιώσιμη αλληλεία σε επίπεδο περιβάλλοντος. Έρχομαι στην τελευταία μου διαφάνεια Μπορεί να ενδιαφέρει αυτό κάπου τα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι εδώ είναι ο αριθμός των μελών μας στην Όσιο 2012. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο με πέντε μοναχα φορείς και από χθε βρισκόμαστε στους 39 φορείς από 13 κράτη-μέλη. Περίπου 20 από αυτούς τους φορείς νομίζω είναι παρόντες σήμερα και παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση και προσπαθούν ε, να ασκήσουν επιρροή στα μέλη του Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. καθώ προχωρά ο χρόνο και εφόσον το Κοινοβούλιο αποκτά όλο και περισσότερε εξουσίε στην απόφαση συγκεκριμένα στα θέματα αλίας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και περισσότερος κοινοβουλευτικό έλεγχο από την πλευρά του Κοινοβουλίου και ήταν ενδιαφέρον ότι παρά το γεγονό ότι ήταν μια δημόσια κρόαση δεν υπήρχε αρκετό χρόνο, αρκετό χώρο μάλλον για να καθίσουν οι πολίτε και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση ίσω έχει παραγωνιστεί λίγα και το θέμα τη αλλία στο παρελθόν, αλλά δεν θα ισχύσει αυτό και για το μέλλον, σα το υπόσχομαι. Και αν είναι κριτήριο αυτό το γράφημα, θα έχουμε πολύ περισσότερου φορεί οι οποίοι θα είναι σε θέση να αρρωγήσουν τα μέλη του Κοινοβουλίου στο μέλλον και να εξασφαλίσουν ότι την χάνει τη πρέπουσα προσοχή το έργο αυτό το οποίο γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν κάλυψα όλο το χρόνο μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκη Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι έχουν κάτσει, δεν υπάρχει κανένα όρθιος από ό,τι βλέπω. Στη συνέχεια για 10 λεπτά ο κύριος Αντώνιο Νάπολη, ο οποίος εκπροσωπεί την Αλία της Σικελίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στην εξέταση των προτάσεων που περιλαμβάνει πράσινη βίβλος για την κοινή ελευτική πολιτική, θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες ε, σκέψεις για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που ε, καθόρισαν τον ε, αλλιευτικό τομέα στη Σικελία και κυρίως ε, τα όσα συμβαίνουν στην λεκάνη της Μεσογείου. Θα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση αποτελεσματική που θα πρέπει να δώσει λύσεις που, στα προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τον τομέα και θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις και όχι επιζήμιες λύσεις τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της ελευτικής προσπάθειας και του περιορισμού της, ε, του στόλου παρά το γεγονός ε, τους, ε, ότι διατέθηκαν μεγάλοι πόροι για το θέμα αυτό, έχουν οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα και σήμερα το 88% των αλληλευτικών αποθεμάτων υποβάλλεται σε πολύ μεγάλη πίεση που, που υπερβαίνει στο επίπεδο της βιωσιμότητας και το 30% είναι κάτω από τα βιολογικά επίπεδα ασφαλείας. Το να συνεχίσουμε λοιπόν ε, να ακολουθούμε τις παλιές μας θέσεις και να θεωρούμε ότι η διαφύλαξη των ε, αλλιευτικών ε, πόρων θα πρέπει να γίνει χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις αρνητικές συνέπειες και λαμβάνουμε υπόψη την αρχή της ε, πρόληψης ε, δεν είναι μια επιλογή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την κοινωνική καταστροφή ε, και την κατάρρευση του αλληλευτικού συστήματος και του στόλου της θα εξακολουθεί να υπερισχύει η θέση ότι η μείωση των πόρων θα πρέπει να, να είναι αποκλειστικά το μέτρο που θα εφαρμόζεται και θεωρούμε ότι ε, αυτό μπορούμε να το θυσιάσουμε. Κανένας δεν μπορεί να δείξει ε, ποιος είναι ο υπεύθυνος ε, και εξακολουθεί ε, να ε, είναι επιζήμιο για την υγεία των ε, θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ε, έχουμε ε, πάρα πολλές μεγάλες μειώσεις πληθυσμού, κυρίως στη λεκάνη της Μεσογείου και υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τον καθαρισμό των λιμάτων. Πολλά από αυτά πηγαίνουν στην θάλασσα και διαταράσσουν την περιεκτικότητα σε άλλα των οικοσυστημάτων. Επίσης, τεράστιες ποσότητες δηλητηρίων, ε, βαρέων μετάλλων, ε, ε, απορρίμματα από την χημική και πετρελοχημική βιομηχανία πέφτουν στην Μεσόγειο θάλασσα, η οποία θεωρείται ο μεγάλος υπόνομος της περιοχής. Και εξαφανίζονται ε, με σκάφη που βυθίζονται τεράστιες ποσότητες ε, χημικών λιμάτων τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Η μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια θεωρείται κατηγορηματική λύση. Οι αλληλείς, ε, οι οποίοι είναι αυτοί που διαστηριοποιούνται στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και δεν τους ρώτησε κανένας για τις επιλογές που θα λάβουν. Ίσα ίσα υποχρεώθηκαν να επιβληθούν ε, να ληφθούν τα μέτρα και τους υποχρέωσαν να μειώσουν τις ημέρες αλίευσης, ε, να αλλάξουν τα αλλιευτικά τους εργαλεία, να μειώσουν τα δίχτυα τους. Δαπανώνται εκατομμύρια ε, ευρώ για να παροπλιστούν σκάφη, να αλλάξουν ε, εργασία οι αλληλείς και δεν έχουν ε, αλλάξει τίποτα. Υπάρχουν μεγάλα πελαγικά ε, σκάφη τα οποία χάνουν τη δουλειά τους από τους στόλους τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν κατάφερε να προχωρήσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη λεκάνη της Μεσογείου και έτσι οι ανταγωνιστές μας ε, μπορούν να πάρουν κεφάλαια αν θέλετε και οι δικές μας επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κλείσουν. Και έτσι έχουμε μια πολιτική η οποία μπορεί να θεωρηθεί κοντόφθαλμη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα για τις ε, ε, αλληλευτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνονται συνεχώς να μειώνουν την προσπάθειά τους και έτσι χάνονται οι δικέ μας αγορέ. Η κοινή αλληλευτική πολιτική, ε, καθώς επίσης και την, ε, η εθνική και περιφερειακή πολιτική του τομέα, ε, χάνεται συνεχώς, ε, εισάγονται πολύ αυστηροί κανόνες, χάνονται σκάφη και τελικά χάνονται ολόκληρε οι επιχειρήσει και οι απασχολούμενε επιχειρήσει αυτέ. Επίση υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί, περιορισμοί στα μεγάλα πελαγικά είδη, ξυφίε, τόνου, ε, και γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι για τον ερυθρό τόνο. Ε, ένα άλλο παράδεξο της κοινοτικής πολιτικής που ποιος ξέρει από ποιες πιέσεις περιβαλλοντικές ε, καθορίζει τα αλλιεύματα του ερυθρού τόνου βάσει εθνικών ποσοστώσεων ενώ οι τρίτες χώρες μπορούν να αλλιεύσουν τεράστιες ποσότητες ενώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε ε, τα αλλιεύματα παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι είναι παρακολούθηση το είδος δεν μας λένε βάσει ποιων επιστημονικών ενδείξεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε βαθιά κρίση και το γεγονός ότι συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία ε, σημαίνει ότι θα υπάρξουν τεράστιε συνέπειες για την απασχόληση και για, σε κοινωνικό επίπεδο για τις επιχειρήσεις. Επίσης, η παραδοσιακή αλληλεία συνήθως ε, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι μπορεί να έχουμε επιπτώσεις για ολόκληρη την οικογένεια. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να παρεύουμε για να αποφύγουμε μια κοινωνική καταστροφή και για να δώσουμε νέες δυνατότητες αλληλείες ε, στις οικογένειες των αλληλείων. Να περάσω τώρα στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι τρεις είναι οι βασικές πτυχές ο αλληλευτικός τομέας πρέπει να συνεισφέρει στην προάσπιση του περιβάλλοντος και αυτό θα πρέπει να προκύψει από μια περιβαλλοντική ε, επιστημονική προσέγγιση και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, αυτά στην έρευνα ε, για την αλληλεία που γίνεται επί τόπου. Τώρα, η προσέγγιση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από προγράμματα οικονομικής υποστήριξης για τα όσους ενδιαφέρονται και για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις οικονομικού και κοινωνικού τύπου. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτές τις αλληλευτικές επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής ε, πολιτικής θα πρέπει να μην είναι πλέον ε, ε, κεντρική, θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσει που έχουμε σε κάθε περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική διάσταση και συζητώντας με όλους τους ενδιαφερομένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τις βασικές αρχές, τα βασικά στοιχεία και από εκεί και πέρα η επιλογή της πορείας και τις διάφορες ιδιαιτερότητες θα πρέπει να εξετάζονται σε τοπικό επίπεδο οι περιβαλλοντικές συνέπειε για τα αλλιευτικά αποθέματα δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των αλλιέων, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να αυξηθούν οι έλεγχοι σε δραστηριότητε και να υπάρχει μια ανθρώπινη προσέγγιση στα οικοσυστήματα, να υπάρχουν μεγαλύτερε κυρώσει για όσους ε, ρηπαίνουν και καταστρέφουν τα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από την επιστημονική έρευνα και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, αλληλεία η οποία θα είναι οικοσυμβατή και βιώσιμη από οικολογικής πλευράς. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται βάσει των απαιτήσεων της αγοράς. αν ρυθμίσουμε την τοπική παραγωγή και υπάρχουν και ε, επισημάνσεις ποιότητες, θα μπορέσουμε να έχουμε μια βελτίωση των αλληλευτικών επιχειρήσεων. Τώρα, Το να έχουμε δυνατότητα να ε, χρησιμοποιούμε το σύστημα ITQ, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο, διότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα είναι διαφεροποιημένα για κάθε περιοχή. Ελοχεύει ο κίνδυνος, εάν χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο μέτρο, να... Ε, πληθεί η επιβίωση μικρών επιχειρήσεων που ε, δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή αλληλεία. Όλα αυτά δεδομένου ότι τους έχει πλήξει και κρίση τα τελευταία χρόνια και μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάσουν τα δικαιώματα λίας ε, με ε, βάση κάποιες προτάσεις χρηματοοικονομικές που θα τους γίνουν. Και όλα αυτά σημαίνει ότι τελικά όλες, όλα αυτά θα καταλήξουν στα χέρια μικρό, ε, λίγων μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από όλα τα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κοινού πόρους αλίας. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει λοιπόν με τα λιευτικά αποθέματα και να λάβουμε υπόψη μας και τις συμφωνίες που υπάρχουν. Μπορεί να εξαντληθούν οι κοινοί πόροι και να μην υπάρχει δυνατότητα να τους προστατεύσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και να υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες προκειμένου να μπορέσουμε να ε, μάθουμε βάσει ποιων μελετών καταλήγουμε στα συμπεράσματα ε, να μειωθεί η αλληλευτική προσπάθεια που για κάποια είδη τα οποία θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Επίσης υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για το αν είναι σωστά τα επιστημονικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους της ε, ανάλογα με το αλληλευτικό είδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ε, η μεγάλη βιομηχανική αλληλεία και η μικρή κλίμακας παραδοσιακή αλληλεία η μεγάλη κλίμακα αλίας ε, είναι μεγάλων διαστάσεων και έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ενώ η παραδοσιακή αλληλεία συνήθως είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και βασίζεται σε χρόνια ε, προσωπικής δουλειάς ε, και τα οικονομικά ωφέλη είναι ελάχιστα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχει το λόγο για 10 λεπτά ο κύριος Οντόναχιαν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλιέων Παραγωγών και πρόεδρος της Νομοσπονδίας Ιρλανδών Αλλιέων. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παρουσιάζω αυτά τα στοιχεία εξ ονόματος της Ομοσπονδίας των Ιρλανδών Αλλιέων και όχι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Αλλιέων σε ό,τι αφορά την ε, Ιρλανδική αλία υπάρχει μια σειρά από κομβικές προτάσεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει και αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε μια σειρά προτάσεων δικών μας προτάσεων σε σχέση με τη μεταρρυθμίση κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Δέκα κύρια στοιχεία έχουμε εντοπίσει σε σχέση με την κοινή αλληλευτική πολιτική από την οπτική γωνία της Ιρλανδικής αλίας. Ξεκινάμε από τους στόχους της Συμφωνίας της Χάγης, τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις, σχετική σταθερότητα, περιφερικοποίηση, επιστημονική έρευνα, αυτοδιαχείριση, ε, αγορά, ικανότητα του στόλου, πρόσβαση και χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να διεξέλθω όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα πιο ουσιαστικά από αυτά τα θέματα. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο μιας κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το να θέσουμε σαφείς στόχου. πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι του οποίου θα εξυπηρετεί αυτή η πολιτική και οι οποίοι θα πρέπει να διαγράφονται με σαφήνεια και να την χάνουν προτεραιότητος. Δεν θεωρούμε, όπω ελέγχθη από τον κύριο Άμστρονγκ, ότι το MSY είναι ένας πραγματικός γενικός στόχος και μπορεί να έρθει και σε σύγκρουση με την διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες για όλους τους εμπλεκόμενους και δεν μπορούμε να έχουμε 625 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αλία αυτή τη στιγμή. Και προφανώς πρέπει να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή των επαγγελματικών κλάδων. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι η Συμφωνία της Χάγης του 1976, η οποία προστατεύει διάφορες περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την αλληλευτική δραστηριότητα και υπάρχουν 17 τέτοιες περιπτώσεις δίνει συγκεκριμένο τονά στην Ιρλανδία και τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί αυτό, αυτή η απόφαση και να ε, ενσωματωθεί σε μια μεταρρυθμισμένη αλληλευτική πολιτική. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει για, από την πλευρά της Ιρλανδικής Αλίας είναι ότι έχουμε μια έλλειψη επαρκούς ποσοστού σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις για τα δικά μας τα νερά της ε, Ιρλανδίας. Νομίζω ότι το διάγραμμα αυτό σας δείχνει ποια είναι η παραγωγικότητα στις ακτές της Ιρλανδίας. Η μεγαλύτερη παραγωγικότητα είναι στο κόκκινο χρώμα, η πιο παραγωγική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο μέρος των αλλιευμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου έρχεται ήδη από αυτή την περιοχή. σε σχέση με τις περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε, μιλάμε για την περιοχή 6 και την περιοχή 7, θα τα δείτε εδώ στο χάρτη. Είναι οι περιοχές ε, γύρω από την Ιρλανδία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το ποσοστό μας. Ήδη έδειξα στο χάρτη ποια είναι η περιοχή η οποία είναι πιο παραγωγική σε ό,τι αφορά την αλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιρλανδική ζώνη σε αυτή την περιοχή είναι 46% της ε, ζώνης 6 και 7. Έχουμε όμως παρόλα αυτά μόνο 16% των συνολικών αλλιευμάτων που προβλέπονται για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδική Αλία θέλει να διατηρήσει μεν τη σχετική σταθερότητα, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια σημαντική τροποποίηση ε, η ποσόστοσή μας για να λάβει υπόψη αυτήν την έλλειψη ισορροπίας. Θεωρούμε ότι η απόφαση της Χάγης που δίνει προτίμηση στις παράκτιες, στα παράκτια κράτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με μια περιφερική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, κοινότητες που εξαρτώνται από την αλία και να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ποσοστώσεις με πιο εφάνταστο τρόπο και οι συμφωνίες ανταλλαγής επίσης με πιο <clears throat> εφάνταστο τρόπο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το σχετικό μερίδιο μας στην αλία. Σε ό,τι αφορά την ε, προσπάθεια αλλιευσή, εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει το μόνο κριτήριο, το μόνο γνώμονα για την αλλιεύση. Δεν υποστηρίζουμε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η αλλιευτική προσπάθεια σαν βασικό κριτήριο. Περιφερικοποίηση και αποκέντρωση. Εμεί υποστηρίζουμε πλήρω μια περιφερειακή προσέγγιση με την προπόθεση ότι η εμβέλεια, η λειτουργία, οι εξουσίες και η λειτουργία αυτή της περιφερειακής προσέγγιση θα πρέπει να είναι σαφής. Δεν θέλουμε μία περιφερικοποίηση που θα οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία και όχι σε αποκεντρωμένες εξουσίες. Πρέπει οι επαγγελματικοί κλάδοι να εμπλέκονται πλήρως στη διαδικασία λήψης απόφασης και όπως έχει ήδη τονιστεί από τον Ιαν Μακκουίν και τον κύριο και επίσης από την οπτική γωνία της Ιλλανδίας θεωρούμε ότι η περιφερικοποίηση και η αποκέντρωση δεν είναι ο κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε πελαγικά είδη, την αλία πελαγικών ειδών. Τέλος, εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενισχυμένος ρόλος για τα περιφερειακά συμβούλια αλίας. Θέλουμε να ενισχυθεί ο συμβουλευτικό τους ρόλος. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιστημονική έρευνα, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα, Θέλουμε στην ε, περίπτωση της επιστημονικής έρευνας που υπήρξε ένα σημείο διαμάχης μεταξύ των εμπλεκομένων και των αλλιέων εδώ για πολλά χρόνια, θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή, η οποία δίδει συμβουλές ε, για τα αλλιεύματα. Δεν πρέπει να συνεχίσει να αγνοεί τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ακόμα και τις κοινωνικές, τις οποίες αγνοεί απόλυτα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πλοίων που αλλιεύουν κάθε μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τη γνώμη, τις γνώσεις που αποκτούν αυτοί οι αλληλείς στις επιστημονικές μας μελέτες και αυτό ίσως γιατί Είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις αξιολογήσεις και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε με ευρύτερο τρόπο πώς θα κάνουμε αυτές τις αξιολογήσεις. Θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους συλλογής δεδομένων λοιπόν και να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το περιθώριο αβεβαιότητας της αξιολογής τις οποίες ε, κάνουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η αβεβαιότητα για πολλά θαλάσσια είδη. Θεωρούμε ότι οι ίδιοι αλληλείς μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο εάν εξασφαλιστεί η ενεργή τους εμπλοκή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, τα προβλήματα αυτά. Νομίζω τώρα ότι έχω καλύψει τα κύρια θέματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θίξω σε σχέση με το ζήτημα αυτό και ίσως μπορώ να κλείσω λέγοντας ότι προφανώς και το θέμα χρηματοδότησης είναι ένα σημαντικό συστατικό οποιασδήποτε κοινή αλληλευτικής πολιτικής και θεωρούμε ότι μια μεταρρυθμισμένη κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να έχει συγκεκριμένε ρήτρε και πρόνοιε σε σχέση με τη χρηματοδότηση όλων των πτυχών τη κοινή αλληλευτική πολιτική και δεν θα πρέπει να εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία και μόνο η χρηματοδότηση αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση και δέσμευση η οποία θα εμπλέκει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Αλίας για να μπορεί να δίδεται η κατάλληλη χρηματοδότηση για όλες τις πτυχές της κοινή αλληλευτικής πολιτικής μεταξύ των οποίων και αυτά τα οποία έχουμε τονίσει εδώ που είναι τα θέματα επιστημονικής έρευνας. Η Ομοσπονδία των Ιρλανδών Αλλιέων θεωρεί ότι έχουμε ενώπιόν μας μια χρυσή ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια λειτουργική κοινή πολιτική αλλίας μετά από το 2013 και εν κατακλείδη θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο δεν έχω αναφέρει ακόμα το θέμα της αγοράς για τα αλληλευτικά προϊόντα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τιμών. Χρειαζόμαστε νέους κανονισμούς αγοράς οι οποίοι δίνουν την απαραίτητη υποστήριξη στους αλληλείς Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις τιμές των προϊόντων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Ντόνοχιου. Ακολουθεί ο κύριος Φεντερίκο Περέιρα από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Αλίας της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να γίνει αυτή η ακρόαση η οποία περιλαμβάνει τους κύριους παράγοντες στον τομέα αυτό και εφοπλιστές και αλληλείς με στόχο να υπάρξει μια ρεαλιστική πολιτική αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω λεπτομεριακά όλο αυτό το σύνολο και το πλέγμα των ερωτήματων, ερωτήματων που τίθενται σε σχέση με τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Θέλω όμω να σταθώ σε τρία θέματα τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω και αποφασιστικά μέσα στην προβληματική αυτή. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι πολλές φορές η συζήτηση επικεντρώνεται στην αηφορία των πόρων και θεωρούμε ότι αυτό είναι το μόνο θέμα. Παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, προφανώς υπάρχει γενικό συμφέρον για την αηφορία, η οποία είναι απαραίτητη για την αηφορία του ίδιου του αλληλευτικού τομέα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πολιτική αλίας μπορεί να αφρωθεί μονάχα σε σχέση με τους πόρους. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπίσουμε ήδη από την αρχή συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους για την πολιτική ε, πολιτική αλληλείας που πρέπει να είναι κατά, κατά, κατά πρώτο λόγο. Η εξασφάλιση τροφοδοσίας σε ηχθείες για ανθρώπινη κατανάλωση με υψηλή ποιότητα και δεύτερον η διατήρηση των πολλαπλών αλληλευτικών κοινοτήτων που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται μόνο από την αλληλεία. Ήδη στο Μάρτιο 2005, σε μια κρόαση αυτή τη Επιτροπή, τονίσαμε ότι ο κύριο στόχο τη αληθικής πολιτική θα πρέπει να είναι η προώθηση του εξυγχρονισμού και τη ανάπτυξη του τομέα, με σεβασμό βέβαια τη απαραίτητη ισορροπία των αλληλευτικών πόρων, με στόχο να εξασφαλίσουμε μια τροφοδοσία σε ποσότητα και ποιότητα του, του κοινού, τη διατήρηση των θέσεων εργασία και τη βελτίωση των συνδικών εργασία και ζωή των αλλιέων ιδίω στι ε, παράκτιε περιοχέ που εξαρτώνται πιο πολύ από την αλεία. Είναι σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που προτείνει η Πράσινη Βίβλο. Μα περιπτώσει είναι μια προσέγγιση η οποία πιστεύουμε ότι <clears throat> αντιμετωπίζει καλύτερα το στόχο μια ευρωπαϊκή πολιτική αλληλεία στον ορίζοντα του 2000. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη διαδικασία λήψη απόφαση. Φυσικά, αυτό αφορά τη διαχείριση των πόρων αλλά και όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα εμπίπτουν στην πολιτική αλία. Σε ό,τι αφορά τους πόρους πιστεύουμε ότι μία διαχείριση σε τοπικό επίπεδο είναι αυτή η οποία προσαρμόζεται καλύτερα στους στόχους και τις αναγκαιότητες του να έχουμε μια αηφόρο και υπεύθυνη αλία. Και φυσικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο ζητά η συνθήκη της Λισαβόνας. Το ότι θα πρέπει όλη η διαχείριση να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας φαίνεται υπερβολικό γιατί οι κύριοι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση αυτών των πόρων είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η διαχείριση όταν δεν είναι γνωστά τα τοπικά δεδομένα για τον αλλιευτικό στόχο, στόλο και τα είδη τα οποία αλληλεύουν. Το να υπάρχει λοιπόν μια τάση να αποκεντρώνει μηχανισμοί του ελέγχου δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να επιβληθεί μια πολιτική η οποία είναι κεντροποιημένη και συγκεντρωτική και δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες των εμπλεκομένων. Το να δοθούν οι αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη και η υποστήριξη στους αλληλείς μέσα από τις οργανώσεις τους και να μπορούν να συμμετέχουν στο βαθμό του δυνατού, αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να δώσουμε μια αποτελεσματική και αηφόρο ε, λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των πόρων. Το τρίτο θέμα είναι το θέμα της πρόσβασης στους αλληλευτικού πόρους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο το 2002 θεωρήθηκε απλώς μια παρέκκληση. Συγκεκριμένα το να κρατηθεί ο χώρος των 12 μιλίων για τους εθνικούς αλληλείς σε κάθε κράτος μέλος. Και μπορεί κανείς να φανταστεί να υπάρξει μια επέκταση στα 24 στα 50 ε, μίλια, ναυτικά μίλια, αντίστοιχα με το, την έκταση των, ε, της υφαλοκρηπίδας και ακόμα και στα 200 μίλια για τις υπερπεριφερικές περιοχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρόσβαση πέραν αυτού θα πρέπει να είναι παγκόσμια και να μην είναι ιδιωτικοποιημένη η θαλάσσιοι πόρη. Επομένω, απορρίπτουμε την δυνατότητα να υπάρχουν μεταφερόμενε ποσοστώσει, γιατί για μα αυτό θα οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση ιδιοκτησία των ε, ποσοστώσεων και του δικαιώματο τη αλίας και σε μια ιδιωτικοποίηση των θαλάσσων τούτων λεχθέντων υπάρχει και μια ένα άλλο σύνολο ερωτημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μερικά από αυτά τα ερωτήματα τίθενται εξάλλου και από την ίδια την Πράσινη Βίβλο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των πόρων, πέραν τη ανάγκη να υπάρξει μια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο αποκεντρωμένη, η οποία αναλαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και τι ιδιαιτερότητε κάθε χώρα και κάθε αλληλευτική περιοχή, κάθε αλληλευτικού στόλου και κάθε αλληλευτικού πόρου, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι αλληλεί στην επίλυση προβλημάτων και στην εκτέλεση των πολιτικών και όλα αυτά να εδράζονται στις επιστημονικές γνώσεις. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και υποστήριξη με ανθρώπινους και υλικούς πόρους στα εργαστήρια μελετών επιστημονικών. Συγχρόνως είναι απαραίτητη η παρουσία των αλλιέων και η χρήση των γνώσεών τους παρά το γεγονός ότι αυτό έχει γίνει εν μέρη από τα ΡΑΚ, από τα κοινά συμβούλια τα συμβουλευτικά αυτά συμβούλια, είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη στην οργάνωση των αλλιέων και στην κατάρτισή του για να επιτραπεί μια καλύτερη συμμετοχή του όχι μόνο στα περιφερειακά συμβούλια, αλλά και στι οργανώσει παραγωγών σε φορεί οι οποίοι μπορούν χάρη στη γνώση του να συμβάλλουν σε μια καλύτερη ε, διαχείριση. Τα τεχνικά μέτρα και τα σχέδια ανάκαμψης μερικά από τα οποία είχαν θετικά αποτελέσματα, θα γίνουν καλύτερα κατανοητά και αποδεκτά όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των αλλιέων στους στόχους αυτούς και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξη προς τους αλλιείς. Μία πολιτική η οποία οδηγεί σε μία τυφλή διαδικασία παροπλισμού πλοίων δεν έχει καμία ικανότητα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα γιατί δεν έχει σαφή κριτήρια τις περισσότερες φορές και αυτό το οποίο λέγεται εφημιστικά προσαρμογή των στόλων αλίευσης δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, αντίθετα οδηγεί σε μια καταστροφή χιλιάδων πλοίων και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Όπως έχει ακολουθηθεί αυτή η πολιτική λοιπόν μέχρι τώρα πρέπει να εγκαταληφθεί. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε τους θαλάσσιους πόρους είναι να εξασφαλιστεί ένα λογικό επίπεδο εισοδημάτων για τους αλείς και τους εφοπλιστές των αλευτικών πλοίων. Το γεγονός ότι έχουν μείνει τελματωμένες οι τιμές στον καταναλωτή, ενώ αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, δεν επιτρέπει ένα αξιοπρεπές εισόδημα και επομένως δεν επιτρέπει στους αλλιές να συνεχίσουν την αλληλευτική δραστηριότητα. Τώρα υπάρχει μια παρέμβαση στην ε, εμπορία με τιμές οι οποίες θα είναι διαμορφωμένες από την παρέμβαση και η συμμετοχή των αλλιέων σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουν να εμπλέκονται σε μηχανισμούς ε, υποστήριξης, όπως προβλέπεται σε άλλες κοινέ οργανώσεις της αγοράς, είναι για μας μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν. Η αξιοποίηση των νυχθείων μέσω από εκστατείες προώθησης και εγγύηση ελαχίστων τιμών πρέπει να είναι κομμάτι μια κοινή πολιτική αλληλεία. Όπω επίση και η υποστήριξη για το κόστο των καυσίμων που είναι θεμελιώδη για τον τομέα αυτό. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη, τα έσοδα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αθέμητη, τις αθέμητες μορφές ανταγωνισμού από τρίτες χώρες που δεν υπακούν στους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις όπως ο αληφτικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να απαγορευτεί εξάλλου δε η εισαγωγή ψαριών από πλοία τα οποία αλλιεύουν με σημεία ευκαιρίες. Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξης στην μικρομεσαία αλία, λαμβάνοντας υπόψη και την πολυμορφία αυτής της αλίας, όχι μονάχα γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό και απαράγραπτο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων που αναφέραμε σε μια πολιτική αλίας, δηλαδή η τροφοδοσία των καταναλωτών με υψηλή ποιότητα αλεία και διατήρηση των αλλιευτικών κοινοτήτων, αλλά επίση είναι και σημαντικό για να διατηρήσει μια υγιή σχέση, σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον του, που αυτό θα πρέπει να είναι και αυτό ένα σημαντικό στόχο για μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια και πριν ξεκινήσει η συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιαννή, πρόεδρο της Λέγκα ε, Πέσκα, που είναι μια ε, ομοσπονδία ε, Ιταλών Αλλιών Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε θα αποφύγουμε συστηματικά να μπούμε σε λεπτομέρειες ως προς την πρόταση γιατί έχουμε το κοινό κείμενο της Ευρωπαίας και Κοζεκά. Το προσυπογράφουμε το κείμενο αυτό. Θα επιμείνουμε λοιπόν αποκλειστικά μόνο στη φιλοσοφία της Πράσινης Βίβλου και σε πράγματα που δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος και δεν μπορούμε λοιπόν να τον αφιερώσουμε σε θέματα για τα οποία συμφωνούμε. Τι δεν μας πείθει λοιπόν. Η ανάλυση της πράσινης βίβλου ξαναπροτείνει παλιά εργαλεία και κλισέ που έβαλαν σε κρίση όλη τον αλληλευτικό κλάδο. Αν οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΛΠ έχουν στόχο να αλλάξουν με βάση μιας αναγνωρισμένης χρεοκοπίας, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπολογίζουμε σε κριτήρια και μεθόδους εσφαλμένες. Ιδιαίτερα τη στιγμή που βλέπουμε μια κατάρρευση οικονομική, εργασιακή, κοινωνική με τα μέτρα αυτά, χωρίς βελτίωση των πόρων. Όξυνση των ελέγχων, ανοχή μηδέν, με μέτρα συχνά πολύ περιστασιακά που ευνόησαν ουσιαστικά την παρανομία. Και όλα αυτά χωρίς υποστήριξη μιας σωστής συνοδευτικής κοινωνικής πολιτικής που εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος παρόν από την Πράσινη Βίβλο. Ναι, να δούμε τα πράγματα ολιστικά όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και ναι, στην ανάγκη μιας μεγαλύτερης ενοποίηση της ΚΑΛΠ με τον ευρύτερο προβληματισμό για τη θάλασσα. Ωστόσο η πράσινη βίβλος δεν είναι αυτό που περιμένει ο κλάδος. Παράλληλα με την υπερεκμετάλλευση δεν αναλύθηκαν όλα τα άλλα προβλήματα έχουν άμεση επίπτωση στη διαθεσιμότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των αποθεμάτων. Η αύξηση της οξύτητας στη θάλασσα, η υπερθέρμανση των ωκεανών, οι αλλαγές στο κλίμα, οι εξορρυκτικές δραστηριότητες, οι θελάσσιες μεταφορές, η διάβρωση των ακτών, οι στρατιωτικές απαγορεύσεις, και παρεμβάσεις όλοι είναι εξωγενείς παράγοντες που αλλάζουν το οικοσύστημα, που βάζουν σε δοκιμασία το θαλάσσιο οικοσύστημα και που έχουν αρνητική επίπτωση στη σταθερότητα των βιολογικών πόρων. Ωστόσο η πράσινη βίβλος δεν τα λαμβάνει υπόψη αυτά στον ισολογισμό που κάνει της οικονομίας και της ε, ε οικολογίας, ε, οικολογίας όσον αφορά τα είδη χθειών. Πρέπει αυτά όλα να καλυφθούν και η μελλοντική ΚΑΛΠ θα πρέπει αποτελεσματικά να λαμβάνει υπόψη τις θεωρίες της οικολογίας που λαμβάνει υπόψη την αρχή της σύνεσης και για τη διαχείριση των πόρων αλλά και για την προστασία στο δικαίωμα εργασίας. Η ανάλυση της πράσινης βίβλου ξεκινάει από ένα ιδανικό σενάριο και περιγράφει με μεγάλη επιπολαιότητα ενάμεσο μέλλον στο οποίο θα έχουμε μια ανθούσα αγορά χάρη στην αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, μια ε, πρωτοποριακή βεδοκαλλιέργεια, μικρό κόστος παραγωγής, εμπορική ικανότητα που θα κάνει τις επιχειρήσεις μας ευημερείς, ισχυρές και καλά αναπτυγμένες. Πολύ συναρπαστική αυτή η προοπτική, αλλά είναι γραμμένη πάνω στην άμμο των κενών λόγων. Είναι μια στάση που δεν σέβεται όσο θα έπρεπε μια κατηγορία που περνάει σοβαρή κρίση. Ασφαλώς μας λείπει το πνεύμα που θα μας επέτρεπε να καταλάβουμε το νόημα. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι αδιαφορούμε γι' αυτό, γιατί το θεωρούμε κακής ποιότητας. Έπειτα, στην ανάλυση της πράσινης βίβλου, στηριζόμαστε μόνο σε μία επιλογή γλωσσική που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ξεπεραστεί. Δηλαδή θέλουμε να βάλουμε την αλία στον εξορρυκτικό τομέα. Αυτή η επιλογή δημιουργεί υποψία, φόβο και δυσπιστία. Η αλία μπαίνει στην πρωτογενή οικονομία. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα τρόπο με εξορρυκτικές δραστηριότητες που αφορά το δευτερογενή τομέα. Εξορίστε το πετρέλαιο, τα ορυκτά, ο χρυσός, τα αδρανή υλικά, τα ψάρια, ψερεύονται, καλλιεργούνται και αντίθετα με τους εξοριξόμενους πόρους είναι ανανεώσιμοι πόροι. Πίσω από αυτό το χοντρό λάθος κρύβεται μια επιθυμία φροηδική να αλλάξουμε την τυπική, το τυπικό φορολογικό χαρακτήρα του πρωτογενού τομέα. Έπειτα η μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ έρχεται σε μια πολύ λεπτή στιγμή της διαδικασίας εκδημοκρατισμού των θεσμικών οργάνων. Άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και είναι θεμητός ο φόβος σχετικά με την αντίσταση που θα προβάλλουν τα κατεστημένα συμφέροντα της γραφειοκρατίας που δεν θέλουν να απαρνηθούν τις θέσεις εξουσίας που έχουν υπέρ μιας διαλεκτικής, πιο συμμετοχικής και πιο δημοκρατικής. Υπάρχουν μερικά χωρία ασαφή στην Πράσινη Βίβλο και συγκεκριμένα μια στάση που διαφαίνεται εκ μέρους των εκπροσώπων της Κομισιόν, πράγμα το οποίο μας ανησυχεί, ότι σαν να θέλουν να νερώσουν, να μετριάσουν κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία συναπόφασης με το άλοθη ότι δεν βοηθάει στο να βρίσκονται λύσεις και ότι καθυστερεί, δημιουργεί χρονοτριβή. Πέραν όμως του, του κλάδου της Αλίας, το Ευρωκοινοβούλιο που μέχρι τώρα είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο, εφεξής γίνεται ένας πυλώνας στην κοινοτική δημοκρατία. Θεμητά, δημοκρατικά, όπως το ψήφισε ο κυρίαρχος λαός και ανεξάρτητο της τις εθνικές Έπειτα μας ανησυχεί και τη στάμπα που βάζει η Κομισιόν προκειμένου μέχρι το Μάιο να έχει ένα σχήμα μεταρρύθμισης σε σχέση με τα μεταβιβάσιμα ατομικά δικαιώματα. Πρόκειται για ένα θέμα που κατ' εμάς χρειάζεται ακόμα βαθιά μελέτη, διότι στη Μεσόγειο αυτή η πρόταση ε, σύντομα θα οδηγήσει σε όρια μη εφαρμοσιμότητα στη Μεσόγειο, το μόνο είδο που υπόκειται σε ποσοστώσει είναι ο κόκκινο τόνο. Στη βιομηχανική αλία προβλέπονται προβλήματα συγκέντρωση των δικαιωμάτων. Μπορούμε να έχουμε και ένα ενδεχόμενο καθεστώς μονοπωλίου. Επομένως η υπόθεση να επεκτείνουμε το καθεστώ των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων και στη μικρή αλία, πέραν από πρόταση, συγγνώμη, αλλά μας φαίνεται η αρχή της ε, μεταβιβασιμότητας θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποκλειστικά στο δικαίωμα της αλίας. Αν δεχτούμε ότι μπορεί μια αλλιευτική άδεια να μετατραπεί σε μεταβιβάσιμο δικαίωμα. Εν πάση περιπτώσει μια τέτοια επιλογή θα είχε καταστροφικές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες για τις ε, τοπικές παράκτειες αλλιευτικές κοινότητες. Το Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη εξέφρασε την επιθυμία στην τελευταία πενταετία και συμφωνούμε κι εμείς την ιδέα του να ενισχυθούν τα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια, να είναι πιο ορατά, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή με το καθεστώς παρατηρητή στα διάφορα θεσμικά όργανα, ξεκινώντας από την Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωκοινοβουλίου μέχρι την Τεχνικο-Επιστημονική Επιτροπή και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Αλίας και Δετοκολιάριας της Κομισιόν και στο Συμβούλιο Υπουργών της Αλίας. Οι νέοι οργανισμοί που πρόκειται να γίνουν δεν θα πρέπει να δημιουργούν επικαλύψεις ε, ή να μειώνουν το ρόλο αυτών των συμβουλευτικών οργάνων. Μάλλον θα έπρεπε να ενισχύουν αυτό το ρόλο αξιοποιώντας διάφορες ικανότητες που υπάρχουν και επαγγελματικές και άλλες. Βέβαια τα κονδύλια είναι πάρα πολύ λίγο. Θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν. Για λόγους σεβασμού της διαφάνειας επίσης θα πρέπει να προστεθούν οι δεσμοί διαχείρισης που μέχρι σήμερα παγώνουν κατά κάποιο τρόπο τη χρήση των κονδυλίων και την ίδια λειτουργία της υποδομής τουλάχιστον όπως συνέφη με το μεσογειακό ΣΕΣΕΡ. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τρεις σύντομες ερωτήσεις σε τρεις από τους ε, ομιλητές. Καταρχάς τον κύριο Μπέρτι Άρμστρονγκ. Είπατε ότι θα θέλετε να γράψει τη σχετική σταθερότητα στα συστήματά μας. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αν αυτό το σύστημα διαχείρισης περάσει μόνο σε περιορισμό αλληλευτικής προσπάθειας, τι θα γίνει. Η δεύτερη ερώτηση. Αν δεν είστε υπέρ του να περάσουμε από τα λιευτικά αποθέσματα στο σύστημα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, ε, της ε, απόδοσης προσπάθειας, πώς θα το κάνετε αυτό, διότι έχουμε αποφασίσει ότι τα όρια αυτά είναι αιτία των απορρίψεων. Και τέλος, τον κύριο Ντόναχιου. Αν το άνοιγμα των ζωνών 6 και 7 γνωρίζετε ότι αν είχε επιπτώσεις ε, στην περιοχή, διότι φαίνεται ότι αυτές είναι οι περιοχές τις οποίες είχαμε τα περισσότερα λιεύματα. Ναι, ευχαριστώ. Η κυρία Λεβί. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να θέσω τρία ερωτήματα. Καταρχήν, στους εκπροσώπους από την Ιρλανδία και την Σκοτία. Αναφερθήκατε στην έννοια του MSC, επικρίνοντας την, δηλαδή την έννοια της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω αν μπορεί κανείς να καθορίσει με καλύτερο τρόπο τη στοχοθεσία και να μην χρησιμοποιεί αυτή την έννοια την οποία επικρίνεται. Επίσης, από αυτούς οι οποίοι έλαβαν τον λόγο, υπήρξαν πολλές επικρίσεις σε σχέση με τον τρόπο που διενεργείται η έρευνα. Θέλετε περισσότερη έρευνα. Ιδίω ο εκπρόσωπο από την Ιρλανδία ζήτησε να υπάρξει μια νέα οργάνωση για μελλοντικέ ε, ερευνητικέ ενέργειες. Αλλά από την άλλη πλευρά πολλές φορές δεν χρησιμοποιούμε πάντα ε, τα πορίσματα των ε, επιστημόνων το συμβούλιο, τα συμβούλια αλίας δεν έχουν πάντα ακολουθήσει τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δώσει οι στατιστικοί, στατιστικές έλευνες. και είναι τεράστια τα ποσά των απορρίψεων. Δεν ξέρω πόσοι τόνοι είναι αυτοί οι οποίοι απορρίπτονται και πάλι στη θάλασσα και έχουμε φυσικά και περιπτώσεις ατασταλιών και απατών ή και καθαρά παράνομης αλίας. Προφανώς λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί η και καθαρα παρανομης αλιες προφανως λοιπον πρεπει να βελτιωθει η ερευνα αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και από την πλευρά των πολιτικών θα πρέπει να υπάρξει και τήρηση αυτών των συμβουλών. Το ερώτημά μου είναι τι θα είχε γίνει αν οι πολιτικοί πράγματι είχαν δεχθεί την, ε, τις εμπειρο... τα πορίσματα τα επιστημονικά. Θα είχε υπάρξει λοιπόν τόσο μεγάλη μείωση των αποθεμάτων γάβρου. Και κάτι ακόμα, το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το ερώτημα η πρόταση της Ocean 2012. Μιλάτε για συλλογικούς πόρους. Φυσικά οι θάλασσες και οι ωκεανοί δεν ανήκουν σε κάποιον. Αν λοιπόν πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτή την κοινή αξία που απαρτίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες, Γιατί όμως δεν θέλουμε να θεσπίσουμε και κριτήρια βιωσιμότητας προηγουμένως πρωτού ανοίξουμε σε όλους την πρόσβαση που να εξασφαλίσουν λοιπόν αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας ότι υπάρχει τήρηση κριτηρίων οικοσυμβατότητος στην αλληλεία και φυσικά να μην καταναλώνεται και να καταδαπανάτε ε, τόση ενέργεια. Ίσως οι, θαϊολευτικοί κλάδοι να το δεχτούν αυτό. Η κυρία Ανδρέας Μπαρέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι για την κυρία Μπελιό. Με εξέπληξε και αν δεν κάνω λάθο κατάλαβα ότι προτιμάτε το σύστημα των τάκ και των ποσοστώσεων. Με εκπλήσει το γεγονός ότι μια οικολογική οργάνωση προτιμά τα τάκ και τις και όχι την αλλιευτική προσπάθεια. Και εδώ προκύπτει η δεύτερη ερώτησή μου. Πώς ε, μπορείτε να προασπίσετε την πολιτική έλλειψη απορρίψεων σε μια πολιτική τάκη ποσοστώσεων. Ο κύριος Ρωμεβαϊρουέδα. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις πολύ γρήγορα. Είναι για διαφόρους εισηγητές και για ένα συγκεκριμένα. Ακούσαμε την έννοια της ανάγκης να ενδυναμώσουμε την παραδοσιακή αλληλεία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος μπορεί να μας δώσει ένα συγκεκριμένο ορισμό για το τι εννοείται με τον όρο παραδοσιακή αλληλεία. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο καθένας από εσάς τον χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο. Για τι περιφέρεια λοιπόν ε, μιλούμε. Δεύτερον, Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης όταν μιλάμε για τη δυνατότητα να ενδυναμώσουμε κάποιες δραστηριότητες, λίγο πολύ αυτό που έλεγε και η συνάδελφος Λεβάν. Ίσως λοιπόν η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε τις καλές πρακτικές. Αντί να έχουμε ασαφή όρια, με ποιον ακριβώ τρόπο θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι όντω αυτή η πρακτική είναι καλή και έτσι να ξέρουμε και ποιος ε, δρά με το σωστό τρόπο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες επισήμανσης και επιστοποίησης για παράδειγμα ε, και ε, κατανοώ ότι αυτό είναι ένα από τα περίπλοκα θέματα και χρειάζονται και κάποιες περαιτέρω σκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξέρω ε, πώς οι διάφοροι εισηγητές θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει επίσης ε, το θέμα της αποκέντρωσης. Το επισημάνατε πολλοί από εσά. Συμφωνώ, κατανοώ ότι είναι πολύ σημαντικό. και όχι μόνο αποκέντρωση προς τις χώρες, αλλά και ίσως και λίγο περαιτέρα. Έχουμε και τις αλλιευτικές ε, δυνατότητες σε διάφορες περιοχές. Μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν να κάνουν με την έννοια του κράτους. Ε, ορισμένες φορές είναι και διακρατικά αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα ε, γιατί ακριβώς ε, περιφερειακή διάσταση μιλάτε. Μιλάμε για περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και να έχουμε εκεί πέρα μεγαλύτερη συμμετοχή ή μιλάμε και για μεγαλύτερη συμμετοχή και να χρησιμοποιήσουμε και τη μέθοδο του από κάτω προς τα πάνω για να συμπεριλάβουμε όχι μόνο και τον ίδιο τον τομέα αλλά και κάποιους άλλους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάτι να πούν ε, ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντα εγώ πηγαίνω έρχομαι μεταξύ δύο επιστροφών και θα το συνεχίσω και σήμερα το απόγευμα. Επομένω έχασα μερικά από τα στοιχεία της συζήτησης αλλά με εκπλήξανε μερικά από τα σχόλια που έχω ακούσει. γιατί διαφέρουν αρκετά από τη δική μου άποψη. Ακούσαμε παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι οι αλληλευτικοί πόροι δεν πρέπει να είναι ο κύριο στόχο τη κοινή αλληλευτική πολιτική και αντίθετα θα πρέπει να ανακαλύψουμε τι ανάγκε τη αγορά και να διατηρήσουμε τι θέσει απασχολήσεω. Αλλά το να πούμε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η αλληλευτική πόρη είναι να λέμε ότι το σπίτι αυτό πρέπει να φαίνεται όμορφο. Αλλά δεν μα νοιάζουν τα θεμελιά του. Χωρί αλληλευτικού πόρου δεν υπάρχει ούτε ε, ούτε ψάρι στην αγορά, ούτε αλής, ούτε τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν η ανάγκη του αυτοπεριορισμού, λέγοντας ότι ακολουθώντας την αγορά. Ανεβαίνουν οι τιμές στην αγορά, οπότε ξεχνάμε τον αυτοπεριορισμό και έχουμε περισσότερα ψάρια. Πάλι πάμε κατά διαόλου. Λέει επίσης ότι θα πρέπει να αποφασίζονται τα αλληλευτικά αποθέματα από τους αλείς. Προφανώς οι επιστήμονες δεν ξέρουν πάντα ποια είναι η πραγματικότητα. Προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα όπως την βλέπουν οι αλλοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνουμε την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και την τροποποιούμε ώστε να μας βολεύει τι ανάγκε μας. Πρέπει οι επιστημονικέ γνώμε να είναι αντικειμενικές από τη φύση του. Ευχαριστώ. Ο κ. Χάπτον. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο γύρος παρεμβάσεων. Μερικά θέματα έρχονται και ξανάρχονται. από κέντρωση. Τώρα μην συνεχίσουμε τη μέθοδο μία λύση για όλους η ίδια. Ο συνάδελφος κύριος Ρωμέβα μας είπε ότι τα αλληλευτικά έθνη ή περιφέρειες δεν είναι το ίδιο με τα κράτη-μέλη. Εγώ προέρχομαι από ένα αλληλευτικό έθνος, τη Σκωτία, που δεν είναι κράτος μέλος αυτή τη στιγμή. Και είπα το πρωί, το ξαναλέω και το έχω πει και στο παρελθόν, ότι θα πρέπει να δώσουμε πραγματική εξουσία για αποφάσεις όσον αφορά την διαχείριση της αλληλείας στα αλληλευτικά έθνη της Ευρώπης. Δεν εννοώ τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μόνο. Βέβαια χρειάζεται ένα ειδικό πλαίσιο και μπορεί ενδεχομένως αυτό να καλύπτει επικράτης δύο διαφορετικών κρατών μελών. Πάμε κάτι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίο ο επίσημος εκπρόσωπος στην Ένωση είναι η Βουλή το 70% της αλληλευτικής δραστηριότητας όμως του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στη Σκοτία και το 20% των αλλιευτικών υδάτων της Ένωσης είναι στη Σκοτία, ανήκουν στη Σκοτία. Γι' αυτό για την αρχή της σχετικής σταθερότητας δεν πρέπει να την απορρίψουμε, διότι είναι λογικό τα αλλιευτικά έθνη που συνεισφέρουν μέσω των πόρων και έχουν συμφέροντα, θα πρέπει να τους εγγυάται κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να δρέπουν τους καρπούς αυτής της δραστηριότητας. Και αυτό αφορά και την διαχείριση, διατήρηση μάλλον των αποθεμάτων. Και έρχομαι τώρα σε μια από τις μεγάλες αποτυχίες της ΚΑΛΠ. Δεν μας έδωσε ένα πλαίσιο που να δίνει κίνητρα στους φορείς να ασκούν αυτή τη διατήρηση. Γιατί τα αλληλευτικά έθνη συγκεκριμένα δεν είναι σαφές ότι θα ωφεληθούν από τις διάφορες θυσίες που προτείνεται να γίνουν. Τι είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε. Στο τέλος της παρέμβασής σας το πρωί για την ίση πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση που είναι ένα από τα βασικά θέματα της ε, μεταρρύθμισης και που είναι ένα πρόσκομα το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε οπωσδήποτε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Άρμστρονγκ σε σχέση με κάτι που είπε. Και ο κύριος Παρέρα επίσης είπε κάτι όταν αναφέρθηκε στο όριο των 12 μιλίων και να επεκταθεί σε 24 ή 50 ή 200. Στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν η Κομισιόν τονίζει ότι σχετικά η διαχειριστική δραστηριότητα ήταν μια από τις σχετικές επιτυχίες της κοινής πολιτικής. Αν τα αλλιευτικά έθνη όμως ελέγχουν τους πόρους για το δικό τους μέλλον, μάλλον καλύτερα θα το πετύχουν παρά ορισμένοι άλλοι που συζητάνε γύρω από ένα τραπέζι και προσπαθούν να βρουν μια λύση, μια που να ισχύει για όλους. Δεν ξέρω αν ο κύριος Άλφσον θα ήθελε να το σχολιάσει αυτό σχετικά με την επέκταση των αποκλειστικών ορίων στη θάλασσα με επικοδομητικό τρόπο. Γιατί αναφέρθηκε στο όραμα και αυτός μιας μεγάλης αποκέντρωσης. Καλύτερα θα είναι να ορίσουμε την αλληλεία μικρού μεγέθους σε περιφερειακό επίπεδο, όπως πρότειναν οι περισσότεροι από εμά. Τώρα, την ενσωμάτωση της αλίας με την ευρύτερη πολιτική για τη θάλασσα. Ο κύριος Γιάννη το ανάφερε αυτό και η συγγήτρια στην έκθεσή της το ανάφερε, στην εισαγωγή της μάλλον. Σας θυμίζω ότι η πράσινη βίβλος της Κομισιόν για τη θαλάσσια πολιτική γενικότερα μας λέει ότι η Ένωση μπορεί και θα έπρεπε να ενισχύσει αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη στη θαλάσσια πολιτική τους. Αυτή είναι μια καλή αρχή να εφαρμοστεί και στο κοινό διαχειριστικό σύστημα για την αλληλεία στο μέλλον. Ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει σήμερα στη συζήτηση και το έκαναν με ένθερμο τρόπο και ειλικρινή τρόπο. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι μια καλόδεκτη εξέλιξη, αλλά αν κάνουμε μια ανασκόπηση στο παρελθόν της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεών τους, Κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένο. Κάποιοι μπορεί να είναι πιο ικανοποιημένοι από τους άλλους, αλλά ποτέ, ακόμα και μια μεταρρύθμιση εκβάθρων δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε εμεί και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν είναι μετά από αυτή τη διαδικασία περνά από την πράσινη βίβλο στη λευκή βίβλο, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι συστάσει οι οποίε θα διατυπωθούν, θα πρέπει να προσπαθήσει να εξέλθει μια ισορροπία και να εξασφαλίσει ότι οι αλληλείς στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά ύδατα και εκτός της Ευρωπαϊκής ε, τα ύδατα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί υπάρχουν χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να παραμείνουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θέλουν φυσικά να μοιράζονται και τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την Νορβηγία, τις νήσους Φαρόες και την Ισλανδία. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια βιώσιμη αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον μιλάμε για ευρωπαϊκά αλληλευτικά αποθέματα. Δεν θέλω λοιπόν να σας καθυστερήσω, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω με τίποτα από όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν από τον Ιρλανδό εκπρόσωπο. Νομίζω ότι έχει καταφέρει να αντικατοπτρίσει πλήρως τις απόψεις όλων αυτών που είναι στον τομέα της αλληλείας στη χώρα μου και των πολιτικών εκπροσώπων της Ιρλανδίας. Πρέπει όμως να αναγνωρίσω και νομίζω ότι αυτό είναι ένας ακρογωνιαίος λήθος για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να υπάρξει και συμμετοχή και περιφερικοποίηση της αλίας. Τα Περιφερειακά Συμβούλια, τα ΡΑΚ, έχουν κρατήσει ένα συμβουλευτικό ρόλο, αλλά μετά από το 2013 θα πρέπει να έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο. Ένα παράδειγμα. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν ξέρουν ότι η έκθεση που είχα σήμερα για το Σαφρίδι αυτή η έκθεση προήλθε από μια διαδικασία εκ των κάτω από τα περιφερειακά συμβούλια. Όλοι μας λοιπόν θέλουμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες διαδικασίες και εξάλλου νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια φόρμουλα μέσα στη μεταρρύθμιση αυτή που να οδηγήσει σε θετικού είδους διάκριση για τα κράτη-μέλη που έχουν τα πιο πλούσια, τους πιο πλούσιους αλληλευτικούς χώρους και σηκώνω το χέρι μου εδώ πέρα ο Σύλλανδος είναι κρίμα να βλέπουμε μερικές φορές ότι έξω από τη δυτική ακτή της Ιλλανδίας εμείς πρέπει να σταματάμε να ψαρεύουμε και ψαρεύουν τα πλοία μόνο άλλων χωρών μελών. Μια θετική λοιπόν διάκριση θα μπορούσε να βοηθήσει μια σειρά από χώρε και θα πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα να ιδιωτικοποιηθεί η αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει εδώ σήμερα έχουν προσφέρει απόψει οι οποίε θα ληφθούν υπόψη και θα μπορέσουμε να ξέρουμε μια ισορροπία, να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις απόψεις και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων να έχουμε βιώσιμη αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο για όλους μας. Ε, ευχαριστώ. κυρία Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Δεν με είχατε δει, γι' αυτό ξαναζήτησα το λόγο. Έχω και εγώ μοναχά τρία σύντομα ερωτήματα, τα οποία αφορούν όλους τους ε, ομιλητές ε, του απογεύματος. Εμένα θα με ενδιέφερε να έχω από την πλευρά των εμπλεκομένων να ξέρω αν μπορούν να προβλέψουν τη δυνατότητα μιας χωροταξία στο θαλάσσιο χώρο, να μπορέσουμε να έχουμε μια οδηγία πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την ε, χωροταξία των παρακτήων περιοχών. Φυσικά θα πρέπει αυτό να εμπλέκει και τους ε, αλληλείς και τους ε, εμπλεκομένους, αλλά το να δώσουμε να αποκεντρώσουμε την αλληλεία με τέτοιο τρόπο ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται μονάχα σε τοπικό επίπεδο, αυτό το βρίσκω επικίνδυνο, δεν θα οδηγήσει σε μια αηφόρο πολιτική. Και επίση το ερώτημα είναι αν είναι επαρκώ κατατισμένη η αλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει περισσότερο στον τομέα αυτό και ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με την ιδέα να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική αλίας η οποία να συνδυάζεται με τις θαλάσσιες μεταφορών, και να αντιμετωπίσουμε το πώς αλληλοεπιδρά χάρη επιδρώνει οι θαλάσσιες μεταφορές με την αλία. Και θέλω να τονίσω λοιπόν αυτά τα θέματα, την αλληλεπίδραση των πολιτικών, την χωροταξία και την κατάρτιση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Όταν μιλάμε για διατηρησιμότητα, νομίζω ότι ο συνάδελφος έχει πολύ δίκιο δεν είναι μόνο διατήρηση των πόρων, είναι και οικονομική και κοινωνική διάσταση. Χωρίς αποθέματα δεν υπάρχει αλία και χωρίς αλίες πάλι δεν υπάρχει αλία. Η αλία είναι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δρά σε ένα πόρο ο οποίο είναι ανανεώσιμο. Πράγμα που δεν συμβαίνει με του ορεικτού πόρου. Θα πρέπει να το προσέχουμε λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να είναι λοιπόν ε, και οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματική. Και ε, έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι το διαπίστωσαν αυτό. Όσον αφορά τώρα στην αλληλευτική προσπάθεια, και εμένα με εξέπλησε η παρέμβαση τη κυρία Μπελιών με την αλληλευτική προσπάθεια και έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι μόνο μέσω τη αλληλευτική προσπάθεια αν έχουμε ένα μέγιστο, μέγιστη βιώσιμη απόδοση ανάλυα και όχι αναείδες μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ε, μειώσουμε και να εξαλείψουμε πλήρως τις απορρίψεις. Γι' αυτό λοιπόν με εκπλήσει και αυτό που λέτε εσείς. Λέτε το αντίθετο και μάλιστα η ελευτική προσπάθεια είναι κάτι το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να ελέγξουμε σε ένα στόλο ε, διότι αυτή τη στιγμή έχουν όλοι δορυφορικό σύστημα ενώ το να έχουμε ε, το άλλο σύστημα το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο δεν θα ήταν και τόσο βιώσιμο. Επίσης, με ενδιαφέρει και το θέμα του οικοσυστήματος. Δεν το ανέφερε κανείς. Στο εγγύς μέλλον θα εστιάσουμε από πλευρά οικο... πλευράς οικοσυστήματος στην Αλία και κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Θα ήθελα να ξέρω και την άποψή σας γι' αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος Περέιρα για τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε την αρχή της ελευθερίας πρόσβασης που βρίσκεται στις συνθήκες, η εκχώρηση αυτή, η παρέκκληση είναι κάτι που μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, διότι κάνουμε αναθεώρηση και μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα πάντα. Εσείς μιλάτε για τη δυνατότητα να φτάσουμε στα 200 μίλια και ούτω καθεξής. Ξέρω ότι κάποιες υπερπεριφερειακές περιοχές το, το ζητούν, αλλά θα πρέπει να είμαστε λογικοί και σε μια κοινή αλληλευτική πολιτική δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων εγώ δεν συμφωνώ. Θα ήθελα να αναφέρω και κάτι που είπαν κάποιοι, το θέμα της υπεραλίευση είναι αδιαφυσβήτητο ότι ένα από τα προβλήματα της ε, κοινοτικής είναι η υπεραλίευση. Ε, διότι αν υπάρχουν υπερβολικές δυνατότητες οδηγούμαστε στην υπεραλίευση και φυσικά ε, όλο αυτό γιατί υπάρχουν σκάφη τα οποία έχουν υπερβολική δυνατότητα αλίευσης. Όλα τα σκάφη βέβαια σε όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα τη υπερβολική δυνατότητα αλίευση. Αυτό ζητάμε και εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ποσοτικοποιηθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να ε, ε, ξέρουμε τι γίνεται. Εάν το γενικεύσουμε δεν το λύνουμε. Θα πρέπει να το ποσοτικοποιήσουμε και αυτό θα πρέπει να γίνει από πλευρά κρατών μιλών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε καν μόνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο από κοινού. Πρέπει απλώ να διαπιστώσουμε ότι όντω υφίσταται πρόβλημα. Ε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Α, ναι, υπάρχει κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος ε, Οντονοχιού. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η επόμενη ε, μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων μπορεί να μην οδηγήσει στην εξαφάνιση του Ταμείου Αλληλείας, αλλά θα έχει λιγότερες δυνατότητες σίγουρα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για θέματα τα οποία είναι ρεαλιστικά. Προσπαθούμε να έχουμε μια λευτική δραστηριότητα η οποία να προσφέρει ένα κάποιο εισόδημα και να είναι ανταγωνιστική. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μα το είπανε πολλοί και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Θα μπορούσε να οδηγήσει και στην αυτοχρηματοδότησή τη. Για τέτοια λεία θέλουμε να μιλούμε στο μέλλον και αυτό θέλουμε να πούμε. Το παρόν σύστημα διαχείριση και διατήρηση των αποθεμάτων είναι σίγουρα ένα μοντέλο το οποίο δεν οδηγεί σε περισσότερο εισόδημα και σε ανταγωνιστικότητα για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν κάνουμε τη μεταρρύθμιση. Θέλουμε να έχουμε ένα αλληλευτικό τομέα ο οποίο θα είναι ανταγωνιστικό, θα δίνει εισόδημα και θα αυτοχρηματοδοτείται. Κατόπιν τούτων να δώσω το λόγο στους ομιλητές, κυρίως αυτούς τους οποίους ετέθησαν ερωτήματα. Όποιος όμως από εσά θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για όσα ακούσαμε, ε, σηκώστε το χεράκι σας και εγώ θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε για αυτή τη συζήτηση 15 λεπτά. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσετε ε, συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Ο κύριος Άμστρονγκ. Σημείωσα τις ερωτήσεις που μου αποφύγθηκαν το θέμα σχετικής σταθερότητας και πώς θα περιορίσουμε την προσπάθεια και αν αυτό θα είναι συμβατό. Θα έλεγα θα είναι συμβατό. Δεν νομίζω ότι είναι ασύμβατη με τον έλεγχο της προσπάθειας μόνο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που δημιουργεί ο περιορισμός της προσπάθειας αν δεν υπάρχει περιορισμός στα αλλιεύματα ή στα αλλιεύματα που βγαίνουν στην ξηρά. Και μένα και το Σόρ μας ρωτήσαν να έχουμε καλύτερες προτάσεις ως προς την αρχή του MSY. Υπάρχουν άλλα δύο κριτήρια, τουλάχιστον. Η μέγιστη οικονομική απόδοση και η μέγιστη κοινωνική απόδοση που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικέ λύσεις. Καλύτερα είναι όμως να προσπίσουμε το σύστημα MSY και δεν είναι πράσπιση του αν πούμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο κύριος Ρομέρα ζήτησε να ορίσουμε την μικρού μεγέθους αλληλεία. Καλύτερη λύση είναι να αφήσουμε κάθε χώρα να το ορίσει, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Τι σημαίνει μικρή αλληλεία στην περιοχή τους και να φροντίσουν για τη διαχείριση αυτή εσωτερικά. Συμφωνώ ότι η αποκέντρωση δεν σημαίνει κατά ανάγκη κράτος μέλος, αλλά περιοχές το στη ακτή της Σκοτίας. Έχουμε τουλάχιστον δύο πρωταγωνιστές εκεί. Σε άλλα μέρη μπορούμε να έχουμε και τέσσερις. Αν θέλουμε λοιπόν αποκεντρωμένη διαχείριση, πρέπει στη, να λάβουμε υπόψη στην περιοχή αυτή της απόψεις τεσσάρων κρατών μελών. Ο κύριος Ντέβις έκανε μερικά άτεγκτα σημεία παρατηρήσεις, αλλά έφυγε. Τα είπε και έφυγε. Ένα με το οποίο δεν συμφωνώ γιατί το είπε δογματικά ότι τα αλλιεύοντα θα παρέχουν προτεραιότητα γιατί άμα δεν έχουμε ψάρια τι θα έχουμε. Έχει δίκιο. Αλλά τι θέλουμε να κάνουμε ένα ενιδρίο με τα, με τα αποθέματα. Βοηθάει αυτό την απασχόληση, βοηθάει τη διατροφή, κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και στοιχεία ως προς τη διατήρηση. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο και οι τρεις αυτές συνιστώσεις όπως είπε σωστά η συγγήτρια. Και οι τρεις συνιστώσεις πρέπει να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια μιας καλής διαχείρισης τα της αλίας. Δεν έχει νόημα να πούμε ποιο είναι πρώτο. Και τα τρία πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη. Από τον Ιαν χάσουν μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα 12 μίλια εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή με βάση την οποία μιλάμε σε σχέση με ένα εκτελεστικό όργανο και ένα μη εκτελεστικό όργανο. Εγώ έχω άμεση εμπορική σχέση, μιλάω μόνο για τα μέλη μου. Μπορείτε εσείς να κάνετε την ερώτηση. Ο κάθε άλλος από πού έχει εντολή, πού στηρίζεται ω προ την εντολή που έχει άλλο αυτό. Τι πάση περιπτώσει για το όριο 6-12 μίλια η Ένωση Τσέζων Αλλιέων θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει για την προστασία του μικρού βιοτεχνικού στόλου πρέπει να μείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Νομίζω απάντησα στα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ κυρία Μπελιών, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολλά τα ερωτήματα που, που τέθηκαν, κυρίως αυτό για τις ποσοστώσεις και τα τάκ έναντι της προσπάθειας και το θέμα των απορρίψεων ηχθείων. Θα απαντήσω εδώ και μετά θα έρθω στο ερώτημα της κυρίας Λέβεν. Νομίζω το κομβικό θέμα, το οποίο πρέπει να απαντήσει η κοινή αλλιευτική πολιτική, είναι ένα πολύ απλό, όχι εύκολο ερώτημα. Πόσο και τι μπορούμε να βγάλουμε από τις θάλασσες, πότε και πώς. Και το τελευταίο ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει αυτό, την αλλιεύση. Το πόσο και τι αυτό είναι ουσιαστικά ένα επιστημονικό θέμα. Και εδώ πρέπει να υπάρξει ένα σύνολο στρατηγικών στόχων μέσα στο οποίο πλαίσιο θα γίνουν αυτέ οι επιστημονικέ έρευνε. Το πλαίσιο όμω θα πρέπει να καθοριστεί από του πολιτικού. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό είναι και ο ρόλο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Όταν λέμε πόσα ψάρια μπορούμε να βγάλουμε από τον ωκεανό, αυτό είναι η θνησιμότητα των ψαριών. Δεν είναι οι εκφορτώσει. Πάντα υπάρχει το θέμα των πιο ασθενών αλληλευτικών πόρων. Γι' αυτό λέμε να εκφορτώνετε όλα τα ψάρια αλλά να τα αφαιρείτε από τις ποσοστώσεις. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τα αλληλευτικά αποθέματα είναι το τι ψαρεύεται, όχι το τι την χάνει εμπορίας. Και εδώ υπήρξε, παραγωγή ένα πρόβλημα με την διαχείριση αλληλευτικής προσπάθειας οι ψάρες μπορεί να είναι πολύ έξυπνοι και αυτό είναι καλό. Πάντα βρίσκουν έναν τρόπο και αυτό μου το λένε οι ίδιοι οι αλληλείς ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να, ψα... να πιάσουμε ό,τι μπορούμε να πιάσουμε μέσα σε μια μέρα και αυτό μας φέρνει πίσω στο θέμα της θνησιμότητος που προέρχεται από την αλία στα αλληλευτικά αποθέματα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο να εξετάσει τα συνολικά αλλιεύματα, ουσιαστικά έχετε να αντιμετωπίσετε τη φαντασία και την εξυπνάδα των αλλιέων που πάντα βρίσκουν τρόπους να πιάσουν πιο πολλά ψάρια. Γι' αυτό στο έγγραφο εργασίας μας εμείς έχουμε προτείνει μια καινοτόμα προσέγγιση για τη διαχείριση η οποία δεν είναι μονάχα με την αλλιευτική προσπάθεια ούτε μόνο με τις ποσοστώσεις, είναι κάπως πολύπλοκη να την εξηγήσουμε, αλλά έχουμε κάνει μια ε, έχουμε κάνει μια προσωμείωση με την οποία μπορούμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα αυτά τα οποία σας παρουσιάζω. Για τα κριτήρια πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια θετική διάκριση υπέρ αυτών οι οποίοι εκπληρώνουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια καθώς και το κριτήριο της συμμόρφωσης. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου καινούριο, μπορεί να είναι καινούριο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα εκδώσουμε ως Ocean 2012 μία έκθεση η οποία εξετάζει 10 μελέτες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου που έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδου συστήματα με θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει από άλλες περιοχές του κόσμου μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Τέλος, για το ερώτημα του κ. Ζότσβικ, το να μεταφέρουμε τα πάντα στις ε, περιφέρειες δεν είναι το καλύτερο. Πρέπει να υπάρχει και κάποιο επίπεδο αποκέντρωσης βέβαια, αλλά η στοχοθεσία για τους στρατηγικούς στόχους και οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση της αλίας θα πρέπει να καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Σοντόνοχιου. Ευχαριστώ. Να απαντήσω συγκεκριμένα σε κάποια από τα θέματα που μετέθησαν. Ο κύριος Στίβενσον αναφέρθηκε στο Ιρλανδικό σύστημα και μου είπε ότι δεν του φάνηκε από τα διαγράμματα που είδε ότι είναι πολύ αποδοτικό. Δεν έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίασή μου. Το είχα στον κατάλογο, αλλά επειδή θεώρησα ότι είχαμε χρονικούς περιορισμούς, θα ασχοληθώ με μόνο πέντε θέματα. Στο διάγραμμα που έβαλα είχαμε την ε, παραγωγικότητα της περιοχής της ε, Ιρλανδίας. Το νέο, η νέα ζώνη αλίευσης της Ιρλανδίας και οι προηγούμενοι ε, έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των. Θα μπορούσα να σας δείξω ένα διάγραμμα που δείχνει την αλλιευτική προσπάθεια και βάσει της προηγούμενης ζώνης αλλίευσης και βάσει της νέας ζώνης αλλίευσης. Και αυτό με οδηγεί να σας πω ότι το νέο, η νέα ζώνη που είναι, πολύ, είναι ένα κουτί πολύ μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι έχει θετικές επιπτώσεις στην ε, παραγωγικότητα της ε, περιοχής. Τώρα, για το δεύτερο θέμα, Νομίζω ότι ο Μπέρτι αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα για το NSY, αλλά εγώ ε, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά εγώ ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Ως βασική αρχή δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στους στόχους. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε μια αντίφαση, διότι δεν είναι δυνατόν να λιεύουμε όλα τα αποθέματα ταυτόχρονα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εμείς κατανοούμε πλήρω ότι υπάρχει η συμφωνία του Ιωάννεσπορκ που σχετίζεται με αυτό. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστέ και να το δούμε αναείδο. Και εγώ έμεινα πάρα πολύ συγκεκριμένο και είπα ότι δεν θα πρέπει να μπει σε ένα στόχο. Θα μπορεί να υπάρχει φυσική αρχή για κάποια θέματα αλλά μάλλον δεν το έχουν πολύ σκεφτεί καλά αυτοί που το λένε για το... και αναφέρονται στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η άλλη ερώτηση ήταν ε, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Νομίζω ο κύριος Ντέιβις έλεγε ότι οι αλληλείς ήθελαν να δημιουργήσουν ε, ε, δικές τους επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που τους βολεύουν. Αν αυτό κατάλαβα από την παρουσίασή μου, μάλλον δεν την είδε πολύ ειλικρινά, διότι αυτό που προσπαθούσα να πω ήταν ότι η παρούσα δομή που λαμβάνουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από τον ISIS, για, κάποιες, ε, για κάποια αποθέματα οι γνωμοδοτήσεις είναι λανθασμένες. Να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα. Το προσφυγάκι είναι το πιο κλασικό. οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αλλάζουν από τη μια χρονιά στην άλλη κατά 40 με 50% κυρίως διότι υπάρχει αβεβαιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πάντα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πλατφόρμα που μας δίνει το εξή. Οι αλληλείς είναι στη θάλασσα κάθε μέρα. Δεν λέω ότι οι αλληλείς γίνονται επιστήμονες. Λέω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε μια μεθοδολογία μέσω της οποίας θα μπορούν οι επιστήμονες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες και να έχουμε μια πιο ακριβή αξιολόγηση της κατάστασης. Σαφώς η βιωσιμότητα των αποθεμάτων είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ο ορισμός για τη μικρή κλίμακα ασαλία που μας ζητήσατε ε, δεν μπορεί να είναι ένας για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει ο Ιταλικός στόλος ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από τον ε, Ιρλανδικό παράκτιο στόλο. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε επί τη βάση κάθε περιφέρειας. Όπως είπε και ο Μπέρτι, ε, θα μπορούσαμε να το δούμε ακόμα και σε επίπεδο κράτου μέλους. Ίσως και αυτό μας κάνει, αλλά μία λύση για όλους, ένας ορισμός για όλους δεν θα ήταν αποτελεσματικό σε αυτή την περίπτωση. Όλοι εμείς υποστηρίζουμε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση και όχι αναπελαγικό είδος αλλά να σας πω το εξής, αν έχουμε αποκεντρωμένη προσέγγιση θα πρέπει να είναι μια κατάλληλη αποκεντρωμένη προσέγγιση, να μην έχουμε μια ακόμα γραφειοκρατική δομή. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε αποκεντρωμένε δομέ, αλλιώ δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Απλά θα δημιουργήσουμε ένα νέο γραφειοκρατικό τέρα, το οποίο ε, θα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη ζωή των Ελληνίων. Νομίζω ότι σπατάλησα αρκετό από το χρόνο που μας δώσατε, κυρία Πρόεδρε, να πω ε, και κάτι όμως για την ε, ολοκληρωμένη πολιτική, θαλάσσια πολιτική. Ναι, μπορείτε, αλλά γρήγορα, γιατί αλλιώς η επόμενη ομάδα ομιλητών ε, θα χρειαστεί να μιλήσει για λιγότερο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ ολοκληρώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω κάτι τελευταίο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Σαφώς θα την υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυτή αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει για τη θαλάσσια πολιτική να δούμε και πάντα βλέπουμε το πώς περιορίζουμε την πολιτική. Θα, ε, θα πρέπει να είναι αμφίδρομη διαδικασία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε υποστηρίζουμε την ε, θαλάσσια ολοκληρωμένη πολιτική, αλλιώς είμαστε κατά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννη Περέρα και Νάπολη παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να περικόψει το χρόνο αγόρευση των υπόλοιπων. Κύριε Γιάννη. Ε, Περέιρα. Ο κύριος Περέιρα, γιατί λείπει ο Γιάννης. Πάρα πολύ γρήγορα κυρία Πρόεδρε να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν του κυρίου Ντέβι. Νομίζω ότι υπήρξε μια πλήρη απάντηση από τον πρόεδρο Λίσανδε και δεν πρόκειται να πω τίποτα περαιτέρω για το πώ καθορίζουμε τι θα πει η βιοτεχνική αλία. Είναι γεγονό ότι υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα, όπω είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, γιατί σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη μας υπάρχει διαφορετικό κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται για το τι είναι βιοτεχνική και μικρή κλίμακο αλία. Το Μάρτιο του 2005 όμως υπήρξε μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό <clears throat> που χαρακτηρίζει πιστεύω πολύ επαρκώς την αλληλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα το κάθε κράτος μέλος όμως θα πρέπει να καθορίσει τι εννοεί με βιοτεχνική αλληλεία. Και τέλος σε σχέση με την σύνδεση αλληλείας και περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφές ότι οι Αλής και η αλία είναι φίλοι του περιβάλλοντος. Είναι καλό για το περιβάλλον να υπάρχει θετική δραστηριότητα αλίας. Και το περιβάλλον είναι φίλος των αλίων. Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των δύο. Η αλία θα πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά ό,τι γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην ίδια την αλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νάπολη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση. Κάποιος αναφέρθηκε στην κοινή επιστημονική μέθοδο για την οποία μίλησα. Σχέση με αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητή μας. Πρόκειται περί του εξής. Οι αλληλείς οφείλουν να συμμετέχουν με τους επιστήμονες στις διάφορες έρευνες έτσι ώστε οδηγίες όπου συνέβη τα τελευταία χρόνια της Ένωσης να μην έχουν σχέση με την πραγματικότητα των αλλιέων άρα και να μην λαμβάνουν υπόψη θεωρώ ότι η ποσόστηση της παράνομης αλλίας το μερίδιο έχει μέσα ένα σκληρό πυρήνα αυτών που επιλέγουν να κάνουν ζημιά στους πόρους σε βάρος τους, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό αλλιέων που δεν δέχονται αυτές τις οδηγίες που τους έρχονται από πάνω. Θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητά τους ως αλλιέων. Άρα τις περιφρονούν, δεν τις εφαρμόζουν. Μια κοινή λοιπόν μέθοδος, μια αποδοχή μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και των αλλιέων θα δώσει καρπούς. Φυσικά ο αλλιέας δεν μπορεί να επηρεάζει, να παρισφρεί στη δραστηριότητα του επιστήμονα, να συμμετέχει, να το λαμβάνει υπόψη. Έτσι δρά και πιο υπεύθυνα, γιατί συμμετέχει στη διαδικασία. Και όλες αυτές οι οδηγίες, το πούμε, που βλέπουν από τις επιστημονικές αυτές έρευνες γίνονται δεκτές με όριμο τρόπο για την βιοτεχνική αλληλεία τώρα. Στην Ιταλία αυτό το ορίζουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη συνιστόσα σε σχέση με το κεφάλαιο που επενδύεται. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Στην έκθεσή μου εγώ αναφέρομαι σε μια ιδιομορφία που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ τότε σε ορισμένες αλλιευτικές μονάδες το ποσοστό της μικρής βιοτεχνικής αλίας που είναι κομμάτι του κοινωνικού ιστού είναι τόσο σημαντικό ώστε πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη, να προστατευτεί στη μεταρρύθμιση έτσι ώστε να μην έχουμε κοινωνική κατάρρευση. Διότι οι επιχειρήσεις της μικρής βιοτεχνικής αλίας χαρακτηρίζονται από τον οικογενειακό τους χαρακτήρα. Μικρή χρήση κεφαλαίου Δουλεύει όλη η οικογένεια. Γι' αυτό η κοινωνική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη όπως πρέπει αυτή την κοινωνική πραγματικότητα και να την προστατεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με αυτό ξεκινούμε το δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Για 10 λεπτά ο κύριος Κώστα Μοντέιρο, διευθυντής του EPMAR από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα το να είμαι εδώ μαζί σας και να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή που γίνεται. Στην συζήτηση αυτή για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής αγοράς με κεντρικό άξονα την πράσινο βίβλο και νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω καταρχήν δύο παρατηρήσεις. Η Πράσινη Βίβλος προχωρεί σε μια αντικειμενική διάγνωση της κατάστασης και μια απεικόνηση κατάστασης όπως ισχύει σήμερα ίσως δεν προχωράει αρκετά στην ανατομή των αιτιών της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι αλευτικές δραστηριότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους λόγους της αποτυχίας της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση εναντί όλων μας που εμπλεκόμαστε στον τομέα της αλλίας. Είναι απαραίτητο να λάβουμε λοιπόν ιδιαίτερα υπόψη τον τομέα της αλίας. Να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο παράγονται οι επιστημονικές γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι κάθε φορά και πιο τεκμηριωμένες, όλο και πιο μακρόπνοης αξίες. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει και μία αλλαγή παραδείγματος στην κοινή αλληλευτική πολιτική για λόγους τους οποίους θα αναπτύξω και να μεταφέρουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής ιδιαίτερη ευθύνη στην επιστημονική έρευνα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να μειώσουμε τα ασφάλματα και τις αβεβαιότητες, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την δύσκολη άσκηση. Εγώ θα ήθελα να επιτρέψω στον εαυτό μου να τονίσει ότι κάποια σημεία είναι πολύ σημαντικά Μερικά άλλα τα οποία ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί από τους άλλους ομιλητές. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά από τα βασικά στοιχεία που έχει η Πράσινη Βίβλος. Κάνει μια διαφοροποίηση καταρχήν μεταξύ της αλίας μικρής και μεγάλης κλίμακος. Εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Το θέμα όμως το, και προφανώς το υποστηρίζω για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς. Γιατί η κάθε μορφή αλίας έχει περιορισμένες ε, περιορισμένους χώρους δράσης πέραν της διαφορετικής συμβολής που έχουν στην τοπική οικονομία και η μικρής κλίμακος οικονομίας υπόκειται και σε συγκρούσεις σε σχέση με την χρήση των παρακτήων χώρων. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Πέραν αυτών όμω, θα πρέπει να καθορίσουμε με σαφήνεια τι είναι η βιοτεχνική αλία, η μικρή κλίμακο αλία για κάθε κράτος μέλος. Δεν έχει την ίδια διάσταση, δεν έχει τους ίδιους λειτουργικούς στόχους σε κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών της ε, βιοτεχνικής και βιομηχανικής ε, και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις γνώσεις ιδιαίτερα στον τομέα της ε, μικρής κλίμακος για να μπορούμε να κάνουμε με υποφελέστερο τρόπο την διάκριση αυτή. Πιστεύω ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη σε ορισμένε περιπτώσεις, σε ορισμένα είδη αλίας, τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σε περιφερειακό επίπεδο. Ενώ σε άλλες μορφές αλίας δεν υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή στην αλία μικρή κλίμακο, ιδίω σε ό,τι αφορά την προστασία των αλληλευτικών πόρων. Χρειάζεται λοιπόν πολλή έρευνα ώστε να μπορέσουμε επί τη βάση επιστημονικών τεκμηριωμένων γνωμών και λειτουργικών αναγκών να καθορίσουμε αυτά τα κριτήρια βάσει των οποίων κάθε χώρα και κάθε γεωγραφική περιοχή θα μπορούσε να εφαρμόσει αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ βιοτεχνική και βιομηχανικής αλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την, την ενσωμάτωση της αλληλευτικής πολιτικής στην θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Έχουμε ένα νέο παράδειγμα. Πώς θα αλληλεπιδρά η αλληλευτική πολιτική με τη θαλάσσια πολιτική γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς συγκεκριμένα η εφαρμογή αυτής της θαλάσσιας πολιτικής θα έχει επιπτώσεις στην αλληλευτική ε, πολιτική. Όπως ξέρουμε, η νέα οδηγία της, ευρωπα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει συγκεκριμένη αντιμετώπιση των θεμάτων περιβάλλοντος στην θαλάσσιες μεταφορές και στην αλία. Και αναφέρονται ορισμένες παράμετροι που είναι ακόμα ασαφείς στη συζήτηση, αλλά εδώ βλέπουμε κάποιους από αυτούς τους ε, παράγοντες εδώ πέρα και εδώ μπορεί να έχουν περιορισμένη ε, επίπτωση στην κοινή αλλιευτική πολιτική σε ό,τι αφορά την προστασία των πόρων. Έχουμε παραδείγματος την βιοπικιλότητα, την προστασία της βιοπικιλότητας. Αλλά όταν έχουμε τροφικές αλυσίδες και όταν έχουμε αλλαγές στην, ε, στο κλίμα που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές ακόμη και καταστροφικές που δεν μπορεί να θεωρηθούν ευθύνη των αλλιέων. Τι θα κάνουμε. Θα έχουμε μια διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα, βάζονται, θα βασίζονται σε δείκτες που έχουν να κάνουν με ένα συνολικό οικοσύστημα. Πώς θα αντιμετωπίσει η πολιτική αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και η αρχή του MSY, της μέγιστης ε, βιώσιμης απόδοσης, να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται σε, όλα τα, σε όλες τις αλευτικές δραστηριότητες. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει η έρευνα να εξασφαλίσει το κατά πόσο η αλληλεία επηρεάζει αυτούς τους δείκτες που θέλουμε να έχουμε σε συνολικό επίπεδο για το περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα στοιχείο λοιπόν της κοινή αλευτικής πολιτικής. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες για τους οποίους η αλληλεία έχει άμεση ευθύνη, άλλοι για τους οποίους η αλληλεία δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση, όπως είναι όπως Ανέφερα προηγουμένω η τροποποίηση των θαλασσίων ρευμάτων, η τροποποίηση του κλίματο, βιομηχανικέ άλλε ανθρωπογενεί επιπτώσει που δεν προέρχονται από την αλία μπορούν να επηρεάσουν ακόμα περισσότερο αυτού του πόρου. Επομένω, η πραγματική πρόκληση σε επίπεδο έρευνα είναι να μπορέσουμε να διακρίνουμε και να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε μια καλύτερη ισορροπία για τους δείκτες αυτούς ώστε να καταλογίσουμε ευθύνες ή όχι στις αλλιευτικές ε, δραστηριότητες και στην ε, ενδεχόμενη βλάβη του περιβάλλοντος. Ένα σχόλιο επίσης σε σχέση με τις δομές διακυβέρνησης που έχουν άμεση σχέση με την ε, έρευνα. Η εμπειρία μας έχει δείξει στην περίπτωση της έρευνας ότι παίζουν ένα πολύ θετικό ρόλο τα, τοπικά, τα περιφερειακά συμβούλια αλίας. Είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για την ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων επειδή έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τα περιφερειακά και τοπικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτικές οι οποίες συνενούν και συνάδουν περισσότερο με τις πολιτικές που ζητούν οι αλευτικοί φορείς και επίσης ευνοούν μια μεγαλύτερη ε, συμμετοχή και ενεργή συμμετοχή στις δομές της διακυβέρνησης της Αλίας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της, ε, των συμβουλών και της διαχείρισης, αυτό μπορεί να μας απασχολήσει για πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να σταθώ μονάχα σε ορισμένα θέματα τα οποία θέτει η Πράσινη Βίβλος. Ιδίως σε ό,τι αφορά το θέμα των μακροχρόνιων στόχων διαχείρισης. Πιστεύω ότι εδώ το MSY είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα εξασφαλίζοντας ε, την ε, το σεβασμό των ε, στόχων του περιβάλλοντος. Τώρα σε ό,τι αφορά την αλία πολλαπλών ειδών και την εφαρμογή του MSY, εδώ θα χρειαστεί να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τα θέματα αυτά. Δεν είναι κατά αναγκή η μόνη λύση η εφαρμογή του συστήματος αυτού. Εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων το οποίο θα είναι μια καλή ενδιάμεση λύση και να έχουμε ποσοστώσεις κατά αλλιευόμενο είδος. Αυτή είναι η μόνη λύση που μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε. Τέλος, το θέμα της υδατοκαλλιέργειας. Μου φαίνεται ότι είναι ένας θεμελιώδης πυ... πυλώνας της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στο, στην πράσινη βίβλο. <clears throat> Πρέπει να είναι σημαντικός πυλώνας της, ε, αλλιε... της ε, πολιτικής. Γιατί αλλιώς θα έχουμε δυσκολία σε ό,τι αφορά τη χωροταξία, εάν δεν λάβουμε υπόψη και την υδατοκαλλιέργεια. Η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θα παίξει ένα αυξανόμενο ρόλο σε ό,τι αφορά την παροχή τροφίμων. Αλλά προφανώς αυτό έχει επιπτώσεις στα παραδοσιακά παράκτια θαλάσσια περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί μαζί με άλλες ε, δραστηριότητες και όχι μόνο την παραδοσιακή αλία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ συγκροωμένων συμφερόντων και αυτό είναι καλό να γίνει και σε επίπεδο πολιτικής ήδη από τώρα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια στιγμή μονάχα, λέει στην Πρόεδρο, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της ε, έρευνας που απαιτεί η υδατοκαλλιέργεια, είναι κάτι το οποίο είναι στρατηγική σημασίας και για την ανθρώπινη ε, διατροφή. Έχουμε τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την διατροφή των ηχθείων, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παθολογιών, σε ό,τι αφορά την πόνη Ευρώπη να αποφύγει να αντιμετωπίσει αυτό το σημαντικό θέμα της καινοτομίας για την υδατοκαλλιέργεια, το θέμα της ε, τροφιμικής ασφάλειας και της πιστοποίησης είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά θέματα και αυτοί οι δύο τομείς της ε, υδατοκαλλιέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοντέιρο. Ο κύριος Πέτερ Μπρίπλινγκ από το Ίδρυμα, από την, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης των Γερμανών Αλίεων. Έχει το λόγο για 10 λεπτά. Meine Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος μιας εθνικής οργάνωσης αλλιέων που είναι απαρτιζόμενη από ενώσεις αλλιέων στην, ε, στη Γερμανία και έχω λοιπόν κατά συνέπεια την τιμή να εκπροσωπώ ένα εκατομμύριο πολιτών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να εξασφαλιστεί μια ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται πολύ πιο έντονα στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της αλίας. Και βλέπουμε ήδη ότι η Κομισιόν ήδη επιζητεί την ενίσχυση των ε, νομοθετικών σας αρμοδιοτήτων παρά το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια καθυστέρηση της λήψης αποφάσεων στον τομέα της αλίας. Και εν μέρη με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν υπονομεύει την ε, απόφαση του Συμβουλίου. Παραδείγματος χάρη το άρθρο 11 λέει ότι τα πλοία αυτά τα οποία ασκούν την αλία βακαλάου στη Βόρεια Θάλασσα θα εξαιρούνται από την προστασία του βακαλάου. Επομένως, μια σειρά από τέτοιες εξαιρέσεις που υπήρξαν στο παρελθόν θα απορρίπτονται στο μέλλον γιατί η Κομισιόν έχει εισαγάγει και πρόσθετα κριτήρια σε σχέση με αυτά τα οποία πρέπει να πράττει μια αλλιευτική δραστηριότητα. αλλά αυτό δεν έχει νόημα να το πράττει η Κομισιόν εάν δεν είναι πραγματικά τεκμηριωμένοι οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτή η λήψη αποφάσεων από την Κομισιόν. Έχουμε πει στον κύριο Φερχόγγεν πολλές φορές ότι δεν θέλουμε να έχουμε μία ε, δικτατορία των τεχνοκρατών στην Αλία, ακόμα και αν είναι πεφωτισμένη. Επίσης, για το θέμα της διατήρησης Τη σχετική σταθερότητα Έχουν λεχθεί πολλά σχετικά, αλλά αν κοιτάξετε πού βρίσκεται η υπεραλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπερβολική ικανότητος αλλιευτικών ε, στόλων, βλέπετε ότι η προσκρούει πάντα η προσπάθεια αντιμετώπισης της ε, υπεραλίευσης από αυτούς οι οποίοι ζητούν εναλλακτικά συστήματα από αυτά των ποσοστώσεων. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ζητούν να τροποποιηθούν οι κατανομές των ποσοστώσεων. Εμείς το απορρίπτουμε και αυτό. Δεν χρειαζόμαστε μια συζήτηση για ανακατανομή, χρειαζόμαστε να έχουμε σαφείς λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Τρίτον, χρειαζόμαστε προφανώς να έχουμε αηφορία, έλεγχο της αηφορίας και επιβολή κυρώσεων αλλά χρειαζόμαστε συγχρόνως να έχουμε και αμοιβέ και θετικά κίνητρα για τους αλληλείς, όταν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν νέες επιδοτήσεις για τις αλληλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες πράγματι λειτουργούν με βάση την αρχή του MSY, γιατί να μην υπάρχει οικολογική πιστοποίηση αυτών των επιχειρήσεων. Αν θέλετε να έχετε αποδοχή των πολιτικών αποφάσεων, θα πρέπει να δώσετε θετικά κίνητρα και στους αλείς και αυτό το θετικό κίνητρο δεν είναι μονάχα το να μην υφίστανται σε κυρώσεις. Ένα δημοκρατικό σύστημα πρέπει να δίνει και, τη, να, και κυρώσεις και αμοιβέ. Τέταρτον, η αλληλεία χάνει όλο και περισσότερο δυνητικούς χώρους αλίευσης από άλλες δραστηριότητες. Οι χώροι της Natura 2000, οι χώροι όπου εγκαθίστανται παραδείγματος χάρη ανεμογεννήτριες κτλ. Στη Γερμανία 40% της αποκλειστικής οικονομικής ε, ζώνης ε, θα καταληφθεί από αιωλικά πάρκα, όπου δεν θα μπορεί να λαμβάνει χώρα αλία. Και επίσης υπάρχουν σημαντικές περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας Natura 2000. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία νομική προστασία για την αλληλευτική δραστηριότητα όταν υπάρχουν νομικές προστασίες για άλλους χρήστες των περιοχών αυτών, ενώ αυτό αφορά μόνο τα αερολικά πάρκα ή την προστασία του περιβάλλοντος. Οι άλλοι δεν έχουν καμία νομική προστασία για τη δραστηριότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για χωροταξία στη θάλασσα, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να καθορίσει νομοθετικά ποια θα είναι αυτή η χωροταξία αφεαυτής. Πέμπτον, χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα. Μας λένε πολλές φορές οι επιστήμονες ότι ορισμένα αποθέματα είναι ουσιαστικά άγνωστα. Πάρα πολλά σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται, πάρα πολλά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα για την ε, ε, παραγωγή ηχθείων είναι άγνωστα. Πάνω από 50% τα 100 των αποθεμάτων είναι σε πολύ μικρό βαθμό γνωστά και δεν έχουμε τη δυνατότητα επί τη βάση αυτών των στοιχείων να αποφασίσουμε σε σχέση με τις αλληλευτικές μεθόδους αν υπάρχει υπεραλίευση ή όχι. 86 <clears throat> λοιπόν τα 100 των υπεραλιευμόνων αυμένων ε, αλλιευμάτων ένα, μονάχα, ένα κομμάτι μονάχα από αυτά καλύπτονται από συνολικά αλλιεύματα. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει μια πρόοδος στην επιστημονική έρευνα σε επίπεδο θαλάσσιας βιολογίας. Θα πρέπει να κάνουμε και μελέτες οικονομικού αντικτύπου και να τις λάβουμε υπόψη. Αν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία σε ό,τι αφορά την θαλάσσια βιολογία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα κριτήρια. Και αυτό σημαίνει περισσότερα μέσα και περισσότερες δυνατότητες σε ερευνητικό επίπεδο. Εκτό και τελευταίο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αλλαγές στο επίπεδο του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Γι' αυτό σας δείχνω και το τελευταίο αυτό, ε, αυτή την τελευταία εικόνα και τα άλλα δεν πρόκειται να τα αναφέρω. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τα θέματα του περιβάλλοντος. Αν θέλουμε να έχουμε υπόψη τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην αλλιευτική πολιτική, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους φυσικούς κινδύνους για τα αλλιευτικά αποθέματα. Να βρούμε τρόπους να μειώσουμε επομένως τους κινδύνους για τα αλλιεύματα. Στην γεωργία θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει παραδείγματος χάρη τη μούχλα στις πατάτες. Αντίστοιχο πρόβλημα όμως είναι η κορμοράνη για τα αλλιευτικά αποθέματα. Για το θέμα αυτό λοιπόν εσείς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήρατε μια σημαντική απόφαση το τελευταίο έτος για να υπάρξει ένα σχέδιο διαχείρισης των κορμοράνων στην Ευρώπη. Και έρχομαι και πάλι στην αρχή της ε, ομιλίας μου. Είδαμε τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος να έχει αρνηθεί να δεχτεί δεσμευτικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτή των κορμοράνων. Σήμερα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην εφαρμογή αυτών των κανόνων για τους κορμοράνους. Η πολιτική περιβάλλοντος στον τομέα της αλίας σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία έχουν να γίνουν σε σχέση με τα προγράμματα Natura 2000. Θα ήθελα να σας ζητήσω εδώ να υπάρχει ένα ισόπεδο γήπεδο σε ό,τι αφορά την Natura 2000 και την αλία εμείς βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τις οδηγίες αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει του Natura 2000 και από αυτό προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αλίας σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η Dogger Bank, παραγματικά χάρη, στην Βόρεια Θάλασσα είναι ένα οικοσύστημα το οποίο το διαμοιράζονται τέσσερα κράτη-μέλη και τα τέσσερα αυτά κράτη-μέλη δεν έχουν ποτέ συμφωνήσει για το τι είναι μια περιοχή αμολόφων και τι όχι. Οι τρει λένε ναι αυτή η περιοχή είναι περιοχή αμολόφων, η τέταρτη λέει ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δυνατότητα να οριοθετήσουμε τις περιοχές αυτές της Natura 2000. Αν δείτε τα στοιχεία αυτά λοιπόν για, τα, ε, για τις περιοχές Natura 2000 στην Ευρώπη θα δείτε πάρα πολλά παραδείγματα αυτής της μορφής. Και κλείνω με μία ε, κατεπίγουσα έκκληση σε όλους να υπάρξει ένα, ισο, ένα ισο, ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, ένα ισόπεδο ε, γήπεδο, γιατί τα επόμενα χρόνια θα δείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η ισότητα στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια για 10 λεπτά ο κύριος Γέρζη Αφαδέρ πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, Μεταποίησης Αλευμάτων της Πολωνίας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καταρχά θα ήθελα να σα. ευχαριστήσω για την πρόσκληση να έρθω εδώ. Είμαι εκπρόσωπο του τομέα τη μεταποίηση ελευμάτων και συνεργάζομαι στενά φυσικά με του αλληλεί. Γνωρίζω πολύ καλά τη θάλασσα τη Βαλτική. Ε, δραστηριοποιούμε στον τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω και πάρα πολύ καλά το θέμα της αλίας στη Βαλτική. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεία θα πρέπει να βασιστεί σε μια σειρά από οικονομικές ε, αρχές. Θα πρέπει να είναι πιο ελαστικά τα σκάφη από οικονομικής πλευράς και θα πρέπει να προσαρμόζονται και στις αλλαγές ε, και στο περιβάλλον αλλά και στις αγοράς. Συμφωνώ λοιπόν με την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτική πολιτικής και αυτό έχει να κάνει και με τις επιδράσεις που μπορεί να έχουμε στη Βαλτική θάλασσα. Στα 10 λεπτά βέβαια που μου δίνονται κυρία Πρόεδρε δεν μπορώ να επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες της Πράσινης Βίβλου και σε όλο το μέλλον της ε, κοινή ελευτική πολιτική. Γι' αυτό ακριβώ θα εστιάσω στα πιο ουσιαστικά θέματα ε, που μας απασχολούν οι επιστημονικέ γνωμοδοτήσει θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στα αλλιεύματα και όχι στι απορρίψει. Το πρόβλημα είναι ότι οι επιστήμονε δεν έχουν πάντα τα επιστημονικά δεδομένα για κάτι τέτοιο και για αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα αποκτήσουν. Είναι σημαντικό τόσο για του επιστήμονε, αλλά και για όσου διαχειρίζονται την αλία και για τον όλο κλάδο. Πρόκειται λοιπόν για μια κοινή επιχείρηση. Με όλα αυτά τα δεδομένα ε, να λείπουν δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοστώσεων των ελευμάτων καθορίζεται από το, Υπουργείο, ε, από το Συμβούλιο Υπουργών Αλληλείας ε, βάσει κάποιων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Αυτό καλό. Αλλά, για παράδειγμα, για το γάδο στη Βαλτική θάλασσα, ο στόχος είναι να έχουμε θνησιμότητα της τάξης ε, το 0,3. Αυτό είναι το επίπεδο και το επίπεδο αυτό το έχουμε επιτύχει φέτος στη Βαλτική θάλασσα. Η ποσόστοση για το γάδο βάσει και των ε, σχεδίων ε, ανάκτησης που έχουμε από τις αρμόδιες επιτροπές, όπως είναι η Επιστημονική Επιτροπή, θα μπορούσε να επιτρέψει να αλλιεύεται μέχρι και τη διπλάσια ποσότητα, αλλά το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε αύξηση μόνο κατά 15%. Πώς μπορούμε να πούμε ότι και πάλι πρόκειται για πολιτική απόφαση η οποία δεν βασίζεται στην επιστημονική βάση και λέει ότι δεν μπορούμε να διπλασιάσουμε τα αλλιεύματα. Όσον αφορά τώρα για τον, ε, τον εξυγχρονισμό του στόλου, ε, να σας πω το εξής. Συμφωνούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ε, ο, το μέγεθος του στόλου δεν επιτρέπει ε, αλληλεία η οποία να είναι αξιαλόγου. Γι' αυτό ακριβώς και μπαίνουμε και στις γκρίζες ζώνες και δεν γίνεται πλήρη δήλωση, πλήρης δήλωση των ελευμάτων. Είμαστε σε μία φάση μείωση των αλευμάτων, αλλά υπάρχει εξή ερώτηση. Ποιο θα είναι το μέλλον του στόλου. Τι στόλο θέλουμε να έχουμε. Η πλειονότητα των σκαφών είναι πάνω των 30 ετών. Και για το 2010 προβλέπεται μία χρηματοδότηση και βοήθεια μέχρι το 40%. αλλά από υπόψη το γεγονός κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, έχουμε τα λεύματα που θέλουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λύση. Δεν βρίσκουμε καμία λύση και τη χρειαζόμαστε την απάντηση. Το θέμα των απορρίψεων τώρα. Υπάρχει ανάγκη να γίνεται ε, επιλογή για τα αλληλεία ε, με παρασυρώμενα δίκτυα. Τα πελαγικά αλλιεύματα του ε, γάβρου, για παράδειγμα, συζητήθηκε ένα αντίστοιχο ζήτημα, αλλά δεν καταλήξαμε σε καμία λύση. Ε, ξέρουμε ότι το θέμα των απορρίψεων είναι σημαντικό και πρέπει να βρούμε μια λύση. Το θέμα των επιρρέψεων σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε και μια ταχεία απάντηση, διότι χάνουμε τεράστιες ποσότητες γάδου και δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο νόημα σε κάτι τέτοιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να ε, βρέχεται κάποιο να πέφτουν στα γόνια του στο κεφάλι του και να λέμε ότι δεν βρέχει. Τώρα, το ITQ. Στην Πράσινη Βίβλο έχουμε μία σειρά από ε, ποσοστώσεις και φαίνεται να υπάρχει μια λογική πορεία για το θέμα της διαχείρισης της αλληλείας και τη δημιουργία κινήτρων για την καλή λειτουργία της ε, αλληλείας. Ε, το ITQ δεν αποτελεί πανάκια για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα. Πέραν από τους βασικούς ε, στόχους υπάρχουν και αρκετές απειλές που προκύπτουν από το σύστημα αυτό και θεωρούμε ότι η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να φεθεί στα κράτη-μέλη. Διότι υπάρχουν διαφορετικά ε, νομικά πλαίσια και διαφορετική αντιμετώπιση για την αλία. Για παράδειγμα, η Πολωνία σκέφτεται να δημιουργήσει συγκεκριμένα μέτρα για την αλληλευτική προσπάθεια από το 2011. Έχουμε λάβει υπόψη μας και το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Δανίας, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε μία σαφή εικόνα ε, και σαφή άποψη μεταξύ των αλλιέων. Ε, η περιφερειοποίηση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Το συζητήσαμε και σήμερα. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αναφέρονται στην πράσινη βίβλο σήμερα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί η διαδικασία λήψη αποφάσεων σήμερα δεν είναι διάφανη. Οι περιφερειακέ οργανώσει αλληλεία παρουσιάζουν την άποψή του, αλλά δεν υπάρχει άμεσο διάλογο μεταξύ των ΡΑΚ, μεταξύ των επιστημονικών συμβουλίων και των ε, κυβερνήσεων. Αυτό το διαπιστώσαμε και τον Οκτώβριο φέτος, αλλά δεν υπήρχε όμως καμία συγκεκριμένη αναφορά στο, προ... πρόβλημα από εκεί και πέρα. Θέλουμε λοιπόν η διαδικασία λήψη αποφάσεων να είναι πιο διάφανη, γι' αυτό και ακριβώ θα πρέπει να συστηθεί μια ομάδα εργασία, δεν ξέρω, η στρογγυλή τράπεζα τη Αλία, τη Βαλτική ε, θάλασσα, όπω είπε παλιότερα ο κ. Βαλάσα, και θα μπορούσαμε να έχουμε εκπροσώπηση από τι περιφερειακέ οργανώσει Αλία, από τον επιστημονικό κλάδο, από του αλληλεί, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλέ φορέ χάνουμε και το θέμα της ε, μεταποίησης. Ε, δεν θα πρέπει να τους παραβλέπουμε. Ε, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ο στόχος του Συμβουλίου λοιπόν θα ήταν να ετοιμάζει συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά συστάσεις σε τεχνικό επίπεδο και έτσι θα μπορούν να λαμβάνονται απο... αποφάσεις κατάλληλες και όχι σαν την αποφάση που, ελήφθηκε για την αύξηση των διαστάσεων των ματιών των δικτών χωρίς να διαβουλευτεί κάποιο στην Περιφερειακή Οργάνωση Ελίας. Ένα ακόμα θέμα, η σχετική σταθερότητα. Η σχετική σταθερότητα θεωρούμε ότι θα πρέπει να μείνει ως έχει. Η διαθροτική πολιτική και η υποστήριξη από τα ε, δημόσιους πόρους. τα διαρθρωτικά ταμεία τα έχει εκμεταλλευτεί ιδεόντω η ελευτική πολιτική και θέλει να συνεχίσει να το κάνει. Στι δημοσιονομικέ προοπτικέ για το 2007-2013 υπάρχουν πάρα πολύ καλέ προοπτικέ ε, για την βελτίωση των υποδομών και θα τι εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Για το μέλλον υπάρχει το θέμα το οποίο σας ανέφερα και πριν, το θέμα του στόλου που γυράσκει και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Αναφέρομαι και στα παλιότερα κράτη-μέλη αυτά είχαν τη δυνατότητα να ανανεώσουν το στόλο του. Τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται και αυτά αυτή την ευκαιρία για να εξυγχρονιστούν και γι' αυτό ακριβώ υπάρχει και το πρόβλημα όπω σα είπα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Πολωνούς Ελληνεί. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώ δεν υπάρχει λύση. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό θα ολοκληρώσω τώρα, κυρία Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στο εμπόριο και στην αγορά. πολλές φορές μιλάμε για τους καταναλωτές. Καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για αυτό που τρώνε. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίησης, μια διαδικασία ανιχνευσιμότητας που θα πηγαίνει από τη θάλασσα μέχρι τον καταναλωτή και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Επιμένω και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό τι μπορούμε να κάνουμε για τις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική και η πολιτική παράπλευρη για τα ε, προϊόντα τα οποία εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δοθεί το πράσινο φως για τα ε, προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η εισαγωγή φιλέτου παγκράσιους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και για τους αλληλείς αλλά και για τους ε, μεταποιητές. Κατευσυγμένα φιλέτα λευκού ε, ψαριού είναι ανταγωνιστικά προς αυτά τα φιλέτα. Μοιάζουν με ψάρια αυτά τα προϊόντα, αλλά τα προϊόντα αυτά έχουν μηδενική διατροφική αξία. Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στον κύριο Εμίλιο Λόρο, Γενικό Γραμματεία της Ένωσης Ελλήνων της Λύρα Καρνότο, για 10 λεπτά. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Για μας είναι ικανοποίηση να μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το πλαίσιο και να δώσουμε και την άποψή μας για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτική. Εκπροσωπώ μια πολύ μικρή κοινότητα αλληλευτική που μπορεί να αποτελέσει σύμβολο της παραδοσιακής αλληλεία στη Γαλλικία θεωρούμε ότι ε, είμαστε εκπρόσωποι της παραδοσιακής αλίας. Ε, κατά την άποψή μας, ε, το, η καταστροφή του, πρεκτή, του Πρεστής, κάτι το οποίο ήταν εξένο προς την καθημερινότητά μας, κατάφερε να κινητοποιήσει τον ίδιο τον αλληλευτικό τομέα για να αντιδράσει από μια εξωτερική απειλή την οποία θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον και θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ε, προοπτικές για την αλληλεία στο μέλλον. Θα ήθελα να επισημάνω λίγο τις πτυχές της παραδοσιακής αλληλείας. Θεωρούμε ότι η παραδοσιακή αλληλεία θα ε, βοηθήσει τους αλληλείς ε, να αναπτύξουν ε, τις δυνατότητές τους. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και ε, είναι εποχιακή αλληλεία, είναι πολύ επιλεκτική και τα αλλιεύματα σχετίζονται πάρα πολύ με τις γνώσεις του αλληλεία, ώστε να ξέρει πότε και πώς θα ρίξει τα δίχτυα του. Στην παραδοσιακή αλληλεία έχει σημασία το σημείο στο οποίο αλλιεύουμε. Επίσης γίνεται κατονομεί πιο ισότιμη των ε, αλλιευμάτων. Πολύ περισσότερα άτομα αποφελούνται από τα αλλιεύματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή αλλίας. Έχουμε την ε, ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Στη Γαλλικία η παραδοσιακή αλληλεία έχει και πολύ μεγάλη κοινωνική σημασία και είναι η μεγαλύτερη πηγή πόρων για τους ε, αλληλείς. Έχουμε περίπου 20.000 άτομα τα οποία απασχολούνται με άμεση απασχόληση και υπάρχουν αλλοίς οι οποίοι αλλιεύουν επί των σκαφών, έχουμε παράκτη αλληλεία και έχουμε περίπου και 5.600 άτομα τα οποία ασχολούνται με την ηχθοκαλλιέργεια. Ε, έχουμε επίσης ολαιόνα και αυξανόμενο ε, αριθμό γυναικών που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αλία στη Γαλλικία είναι ένας από τους βασικούς ε, πόρους ε, ε, στην περιοχή και βοηθάει επίσης και τη λειτουργία σε πολλών άλλων οικονομικών φορέων από αιώνε εκπροσωπούμε τον ε, ναυτιλιακό και αλληλευτικό τομέα της ε, περιοχής και ε, ασχολούμαστε με πάρα πολλέ πτυχέ ανάπτυξης από την κατάρτιση μέχρι και τη ρύθμιση και την εκμετάλλευση των πόρων. Ε, πρόκειται για τους αντιπροσωπευτικούς παράγοντες της, του παραδοσιακού τομέα ή της μικρής κλίμακας αλίας στις ακτές. Εάν ε, υπάρξει κάποιος κίνδυνος για το περιβάλλον πάντα θα πρέπει ε, να οφείλεται στην κακή διαχείριση των πόρων και εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε οικολογικούς, κοινωνικούς και ε, οικονομικούς στόχους για τη βελτίωση. Η παραδοσιακή αλληλεία θα πρέπει να έχει διαφοροποιημένο καθεστώς διαχείρισης για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και βιώσιμη ανάπτυξη στην αλληλεία. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε μόνοι τα προβλήματα και να, αν θεωρηθεί ότι κάποιο τομέα θα πρέπει να μειώσει την ε, προσπάθειά του, οι άλλοι να μην, μπορούν να, ε, μην πρέπει να χάσουν αντίστοιχα τι δικέ του δυνατότητε. Επίση, μα φαίνεται ε, πολύ σωστή η πρόταση της, των 12 μιλίων για τα εθνικά χωρικά είδετα, αν και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύει μόνο για την παραδοσιακή αλληλεία. Τώρα, όσον αφορά τις, ε, τη βοήθεια στην υποδομή, εδώ θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη οικονομική προσέγγιση, δημόσια χρηματοδότηση και θα πρέπει να σκεφτούμε και την ε, ενεργειακή απόδοση των ε, σκαφών και την κατανάλωση καυσίμου που έχουν. οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην, ε, ε, πολιτική, στην αλληλευτική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επενδύσεων, δημιουργούνται προβλήματα, δεν υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας, εργονομίας ε, και κατάλληλης οικονομίας. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία υποτίθεται ότι θα έχει ένα σύστημα κοινωνική προστασία, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπει ε, στους αλληλήσεις να ζήσουν ε, με κατάλληλες συνθήκε. Έχουμε κυρίω παραδοσιακέ επιχειρήσει, οι οποίες ε, κατά πάσα ε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αυτόνομες ή μικροεπιχειρήσεις και η ανάγκη να μπορέσουμε να αγοράσουμε νέα σκάφη για να έχουμε καινούρια ε, δυνατότητες αλληλείας είναι απαραίτητη για να έχουμε αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας. Καταδικάζεται δυστυχώς ο αλευτικός στόλος ε, στη γύρανση και αυτό σημαίνει ότι ορισμένες φορές εγκαταλείπεται η οικογενειακή μορφή παραδοσιακής αλίας διότι κανένα αλίας δεν προτείνει στα παιδιά του που ε, τη σήμερον ημέρα έχουν σπουδάσει και όλα στο πανεπιστήμιο να συνεχίσουν την ε, οικογενειακή επιχείρηση. Ε, ουσιαστικά προάγεται μία αρνητική επιλογή ε, και τελικά αλλιεύει μόνο αυτός που δεν έχει άλλη λύση. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητα επιβίωσης και δυστυχώς αυτές περικόπτονται. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η παραδοσιακή αλληλεία ουσιαστικά ε, είναι ο φορέας που επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς να ψαρεύουμε και δεν θα πρέπει να εξαφανιστούν οι πιο σημαντικοί εκπρόσωποι της. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα ε, για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί κάποιο τι δραστηριότητε τους για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα για την παραδοσιακή αλία. Χρειαζόμαστε μέτρα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και δραστηριότητες διαφοροποίησης συμπληρωματική, όπως είναι η αλία, όπως είναι για παράδειγμα η τουριστική αλεία από την οποία μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικού πόρου. Επίσης θα πρέπει να δουν δυνατότητες ε, για αυτούς οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιώσουν την αλληλεία και να ε, δημιουργήσουν μια πιο βιώσιμη αλληλεία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει συνεργασία με τον επιστημονικό τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συμμαχίε. Να σας πω εδώ ότι υπάρχει ε, συνεργασία με την ΒΒΕΦ και με το Ίδρυμα Longsanet και που πρόκειται για ε, μέτρα για τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα της αλίας. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με το πώς έχει η αλλιευτική δραστηριότητα στη Γαλλικία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα ελλειπούς εμπορευματοποίησης των ε, προϊόντων της. Θεωρούμε ότι υπάρχει άνηση συμπεριφορά σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία έρχονται από εισαγωγή και απαιτούμε τα εισαγόμενα αλληλευτικά προϊόντα να περνούν από τους ίδιους εξαντλητικούς ελέγχους που περνούν τα προϊόντα τα οποία λεύονται από το δικό μας στόλα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται ε, κατανάλωση ελευμάτων τα οποία προκύπτουν από βιώσιμη αλληλεία. Αν θέλουμε να ενσωματώσουμε περισσότερο τις γυναίκες θα πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας ε, όπου αυτή τη στιγμή αποκλείονται οι καθημερινοί οι αλληλείς οι οποίοι ασχολούνται σε παραδοσιακό επίπεδο με την αλληλεία. Επίσης έχουμε προστατευόμενες περιοχές ε, και περιοχές ε, οι οποίες θα πρέπει ε, να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γόνου και αυτές θα πρέπει να γίνονται σε κοινή συνδιαχείριση με τους αλληλείς. Θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες διαφοροποίησης που σχετίζονται με την αλληλευτική δραστηριότητα διότι μπορούν να διαρματρήσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της αλληλείας και θα πρέπει να δημιουργηθούν βοήθειες για την διατήρηση και να δούμε τι γίνεται με την ε, διατήρηση της αλληλείας και να μην χάσουμε μεγάλες κοινότητες αλληλείας. Ολοκληρώνοντας να πω ότι η παραδοσιακή αλληλεία θα επιβιώσει αν λάβουμε υπόψη μας τη σχέση που μπορεί να υπάρχει με την παραδοσιακή αλληλεία στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δίνοντάς τη στο κατάλληλο πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε Λάουρε. Τέλος ο κύριος Μπράιον Οριόρταν, γραμματέας του ICSF. 10 λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελευταίος ομιλητή, αλλά ελπίζω εξίσου σημαντικό όσο μπορώ να ισχυριστώ, να αναφερθώ σε μικρού μεγέθους Αγγλία, βιοτεχνικού χαρακτήρα, μερικές φορές στην ανοιχτή θάλασσα, μερικές παράκτιες, αλλά με γερή κοινωνική βάση και με δεσμούς με που εξαρτώνται από την αλληλευτική δραστηριότητα. Η οργάνωση την οποία εκπροσωπώ, ICSF, τα αρχικά της, ιδιαίτερα ασχολείται με μικρού μεγέθους αλληλεία. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε διεθνείς δραστηριότητες που δημιούργησαν ομαδοποιήσεις μικρών αλλιέων από όλο τον κόσμο, από πέντε υπήρου. Προκειμένου να πάρουμε θέση για τα δικαιώματα και ευθύνε των μικρών αλλιών σε όλε τις χώρες. Στην Ένωση αργήσαμε κάπως να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του είδους της αλλίας. Ελπίζουμε η πράσινη βίβλος στη διαφοροποιημένη μέθοδο και προσέγγιση της να είναι κάτι θετικό. Τουλάχιστον εμεί έτσι το βλέπουμε. Και αυτό που ήταν εμπόδιο στο παρελθόν να έχουμε υπεύθυνου αλλιεί στην Ευρώπη να μετατραπεί σε ευκαιρία. Αυτό ήταν το πόρισμα ενός σεμιναρίου που έκανε η οργάνωσή μας πριν από δύο μήνες ειδικά για τη μικρού μεγέθου και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Για να φέρω κατά λέξη από το, την εισαγωγή των πορισμάτων του σεμιναρίου, οι συμμέτοχοι από 7 διαφορετικές χώρες της Ένωσης, 70 περίπου άτομα συμμετείχαν, συμφώνησαν ότι ο κλάδος μας μπορεί να είναι βιώσιμος και με πολλά υποσχόμενο μέλλον αν του δοθούν αν τύχει μιας δίκης μεταχείρισης και αναγνώρισης. Θα σας πω δύο-τρία λόγια για τα πορίσματα του σεμιναρίου. Σε έξι σημεία. Η μικρού μεγέθους αλία και οι συναφείς κοινότητες και η οικολογική βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων απαιτεί δικαιοσύνη καταρχήν. Καταρχήν οι αλληλείς και αλληλευτικές κοινότητες που εξαρτώνται από τη βιοτεχνική αλληλεία πρέπει να έχουν δίκαιη μεταχείριση στα δικαιώματα πρόσβασης στους πόρους, στις υπηρεσίες, στην πληροφόρηση, στο πώς παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Οργανώσεις μικρής αλίας δεν αναγνωρίζονται από την συστήματα οργάνωσης παραγωγών και άλλα της Ένωσης στη διαδικασία, τη συμβουλευτική και της λήψης των αποφάσεων. Εμείς θεωρούμε ότι οι οργανώσεις και άλλες ενώσεις που εκπροσωπούν τους μικρής αλληλείς θα πρέπει να έχουν και αυτοί ισότιμη πρόσβαση σε αλληλευτικά δικαιώματα και σε ποσοστώσεις και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση με οργανώσεις παραγωγών και άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν μεγάλες αλληλευτικές μονάδες. Δεύτερον, οι διαφορές και ο εντόπιος χαρακτήρας των αλληλευτικών κοινοτήτων. Οι διαφορές είναι βασικό χαρακτηριστικό της βιοτεχνικής αλληλείας και είναι και η δύναμή της κατά κάποιο τρόπο. Αν θέλουμε να ορίσουμε την μικρή αλληλεία παγκόσμια θα χάσουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο ορισμός της μικρής αλληλείας θα πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο, να στηρίζεται στην αρχή της επικορικότητας και πρέπει να δούμε όχι μόνο το μέγεθος και την ισχύ του σκάφους, αλλά τι δεσμούς έχει με την ντόπια κοινότητα, τη δομή της ε, αλλιευτικής μονάδας. Πόση δουλειά χρειάζεται για αυτούς που δουλεύουν στις επιχειρήσεις. Η χρήση της ενέργειας, επιλεκτική αλληλεία και επίπτωση στο περιβάλλον επίσης. Τρίτο, πρέπει να γνωρίσουμε και να σεβόμαστε τις γυναίκες, διότι η μικρή αλληλεία είναι στην οχρά κοιλίδα των πολιτικών της Ένωσης και οι γυναίκες βρίσκονται δύο φορές στην οχρά κοιλίδα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί στη νέα ΚΑΛΠ ο ρόλος των γυναικών ως συνεργαζομένων συζύγων, ως οικονομικών φορέων ανεξάρτητων και η σημασία που έχουν στην κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα της κοινότητας πρέπει να αναγνωριστούν. Τέσσερα, τα δικαιώματα αυτών που δουλεύουν στην βιοτεχνική αλληλεία. Πρέπει να οριστούν και να προασπιστούν, που σημαίνει να ορίσουμε ποια είναι τα δικαιώματα των αλλιέων και των κοινοτήτων τους. Και τα δικαιώματα αυτά να μεταφραστούν σε νόμο, σε ισότιμη βάση με τα δικαιώματα όλων των άλλων. Όταν εγκρίνονται πολιτικές που στηρίζονται σε δικαιώματα για τη διαχείριση της μικρής αλίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συλλογική φύση και η ευημερία, η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτιστική διάσταση. Οπότε εργαλεία διαχείρισης για τη μικρή αλία που προωθούν τα δικαιώματα των ατόμων σε βάρος των συλλογικών συμφερόντων, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την κατανομή σε θέματα αγοράς πρέπει να αποφεύγονται. Η λογική των εργαλείων όπως τα ITC ατομικά μεταφερόμενες ποσοστώσεις με την βιοτεχνική αλία δεν είναι συμβατά. Ας διδαχτούμε από το σύστημα αυτό των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων από άλλα μέρη όπως η Ισλανδία, όπως η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας που αναφέρθηκε ήδη και τα στρεβλωμένα αποτελέσματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας αλλιέων που δουλεύουν στον κλάδο της μικρής αλλίας. Έπειτα με ένα τέτοιο σύστημα η υπεραλίευση και υπερβάλλον στο δεν πρέπει να μπουν από την πίσω πόρτα. Στην περίπτωση της Ισλανδίας υπάρχουν παραδείγματα όπου επετράπει υπερβάλλον δυναμικό στο στόλο μέσω προνομίων που δόθηκαν ιδιαίτερα στις τράτες. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πέμπτο, στη διαφοροποιημένη προσέγγιση, αυτό πρέπει να γίνει και ως προς τη διαχείριση και τα ρυθμιστικά προβλήματα όλων των τομέων. Η ανάγκη μείωση του υπερδυναμικού σε ένα τομέα δεν πρέπει να οδηγήσει σε απώλεια απασχόλησης ή ευκαιριών αλλιεύσης σε πιο βιώσιμους τομείς. Οπότε η αρχή της επικορικότητας θα πρέπει να ισχύει στη διαχείριση της μικρής αλίας και συμφωνούμε με άλλους ομιλητές που το τόνισαν ότι η εθνική διαχείριση, η περιφερειακή διαχείριση μπορεί να στηρίζεται και σε διασυνοριακή διαχείριση. Σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Λύρα υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα διαχείρισης με βάση κοινότητες στη Βόρεια Ισπανία που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και τέλος, το να ληφθεί υπόψη ο τροτός χαρακτήρας και η δυνατότητα ανάκαμψης. Δηλαδή, υπάρχει μια εγγενής, ε, εγγενές στοιχείο εύθραυστου, αλλά ταυτόχρονα και αναπήδησης οικονομικής στις μονάδες αυτές με διαφοροποίηση μέσω προγραμμάτων που να στηρίζονται στην τοπική πραγματικότητα, την ικανότητα αλλαγής, την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να προωθούνται. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, προτείνω η Ένωση να γκρίνει ένα πιο ηθικό πλαίσιο για την ΚΑΛΠ. Μια ηθική πηξίδα που θα κατευθύνει τη μεταρρύθμιση με βάση τη δικαιοσύνη, ίση μεταχείριση, συνετή προσέγγιση, οικοσυστημική προσέγγιση, όπου να λαμβάνονται υπόψη και ο ανθρώπινος παράγων. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε ο Ριόρνταν. Είναι η πρώτη φορά που με αποκάλεσαν Λέδη Πρόεδρε και νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με τη συζήτηση. Έχω έξι άτομα τα οποία θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχουμε μισή ώρα συζήτηση. Ο κύριος Στίβενσον πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Λέδη Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ο Δόκτωρ Μπρέκλιν είναι αυτός ο οποίος έθιξε το σημείο αυτό στην παρουσίασή του, που είχε κάποια απήχηση σε μένα όταν είπε ότι η Γερμανία που δεν ψαρεύει ουσιαστικά καθόλου μπακαλιάρο, ε, δεν, καθόλου γάδο μάλλον, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλεία του γάδου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε στο δυτικό τμήμα της Σκοτίας για αυτούς οι οποίοι δεν ε, πιάνουν καθόλου γαρίδες και παρόλα αυτά δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το σχέδιο ανάκαμψης του γάδου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια λοιπόν, αλλά πρέπει να, να μην ξεχνάμε ότι οι νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα αναδυθούν από όλες αυτές τις συζητήσεις δεν θα διατυπωθούν παρά μόνο δύο χρόνια από σήμερα. Έχουμε μια κοινότητα αλλιέων που βρίσκεται σε ύφεση, που αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος πετρελαίου, αντιμετωπίζει τιμές οι οποίες <clears throat> μειώνονται για τα προϊόντα τους και θα πρέπει να επιβιώσουν τα επόμενα δύο χρόνια. Ελπίζω να με ακούει η Κομισιόν, ελπίζω να σημειώνει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε εξαιρέσεις τις οποίες κανείς δεν μπορεί να επιτύχει. Λόγω των τεραστίων εμποδίων και των αυστηρών κριτηρίων που εμποδίσουν την επίτευξη όλων αυτών των στόχων που περιλαμβάνονται στι εξαιρεσει. Απλώ λοιπόν θα ευχαριστήσω τον δόκτωρα Μπρέκλεν που έφεξε αυτό το ζήτημα και ελπίζω ότι η Κομισιόν το έχει καταγράψει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκρομπάρτσικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριο Σαφάντερ είπε ότι υπάρχει μια ειδική ένωση, μια αλυσίδα κατά κάποιο τρόπο που συνδέει τους ε, αλείς με τους μεταποιητές και τους εμπόρους. Στην περίπτωση Βαλτικής όμως τα πράγματα φαίνονται είναι κάπως διαφορετικά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς προωθούμε την περιφερειοποίηση, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη Βαλτική όπως και τις άλλες θάλασσες. Αυτή λοιπόν η σύνδεση που αναφέρατε, αυτή η σύνδεση έχει να κάνει ουσιαστικά με τη βιομηχανική αλία. Έτσι δεν είναι στη Βαλτική. Ένα δεύτερο ερώτημα. Αναφερθήκατε στην πολιτική απορρίψεων. Εγώ θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο καλύτερα την πολιτική αυτή μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο από την πλευρά της βιομηχανικής αλίας και πάλι για τις ε, απόρριψεις λοιπόν πως μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο κυρία ε, Μπαρέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχάς θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της γερμανικής αντιπροσωπείας Αλίας. Δεν τον βλέπω βέβαια εδώ, αλλά μιλούσε για την υπερβολική δυνατότητα αλίευσης του στόλου και σήμερα το πρωί ε, συζητούσαμε το ενδεχόμενο να γίνει μία κρόση διότι δεν ε, είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ίσως θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Στον εκπρόσωπο της Πολωνίας για την Βαλτική θάλασσα μιλήσατε για την πολιτική απορρίψεων, ε, το έχετε αξιολογήσει, θεωρείτε ότι υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις. Και τέλος ο κύριος ε, Λόουρο, ο Ισπανός εκπρόσωπος από την παραδοσιακή αλία για τη Γαλλικία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί δώσατε ανθρώπινο πρόσωπο στην αλία όπως και ο τελευταίος μιλητής και να σας ευχαριστήσω όπως και στον τελευταίο μιλητή που αναφερθήκατε στο θέμα των γυναικών. Γιατί σε όλη τη συνεδρία σήμερα από τις 9 το πρωί δεν αναφέρθηκε κανείς στη συμμετοχή των γυναικών που είναι τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική και βρίσκεται και στο επίκεντρο της χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην μελλοντική κοινή ελευτική ε, αλληλευτική πολιτική. Μιλάμε για τα θαλασσινά μόνο, όχι ε, για τις γυναίκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου παρέμβαση έχει ως στόχο να επισημάνει κάποια από τα πράγματα τα οποία ακούσαμε εδώ, διότι πραγματικά η παραδοσιακή αλληλεία δεν μπορεί να είναι ο φτωχό συγγενή στην κοινιαλιστική πολιτική, διότι είναι αυτή η οποία συγκεντρώνει του περισσότερου ανθρώπου, ε, επηρεάζει περισσότερο τι ακτέ μα και την, ε, το βιωτικό μα επίπεδο. Όπως και στην ε, γεωργία, ξεκινούμε με την ιδέα ότι είναι οι θεματοφύλακες του περιβάλλοντος η γεωργοί. Με τον ίδιο τρόπο και οι αλληλείς στηρούν αυτή την προϋπόθεση στον τομέα της αλληλείας, διότι έχουμε ανάπτυξη της υπαίθρου και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κοινή αλληλευτική πολιτική και την παραδοσιακή αλληλεία. Κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν για τη διαφοροποιημένη πολιτική, για, τον, ε, για τη μικρή κλίμακα αλληλεία με διαφοροποιημένη ε, βοήθεια και για τα θαλασσινά, εμένα μου φαίνεται πραγματικά πολύ σημαντικό και αν πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι περαιτέρω, θα ήθελα να ξέρω τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε εσείς όταν έχετε προβλήματα, ας πούμε, με την αύξηση των καυσίμων. Και τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε μια βελτίωση για το τομέα της ε, παραδοσιακής αλίας. Έχω κι εγώ ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Μπρέκλιν, η κυρία Λέβιν. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο απευθύνεται στον κύριο Μουντέιρο. Μας μίλησε για την έννοια της ε, μέγιστης βιώσιμης ε, απόδοσης στην περίπτωση μεικτή αλίας, αλίας πολλαπλών ειδών. Τι σημαίνει αυτό σε επιστημονικό επίπεδο, επίση για τον κύριο Μπρέκλιν, ο οποίο δυστυχώ δεν βρίσκεται πια στην αίθουσα. Μας είπε ο κύριος Πρέκλεν για άλλες δραστηριότητες όπως είναι η, τα αιωλικά πάρκα ή το, τα προγράμματα όπως το Natura 2000 που είναι ανταγωνιστικά προς την αλία. Για το Natura 2000 μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό είναι μια δραστηριότητα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση αν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη θάλασσα σαν να είναι απλώς ένα ενιδρίο. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που έλεγε ποια είναι η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακος που απορροφάται από τους ωκεανούς. Και αυτό το οποίο συνιστούσε είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την αποκατάσταση των παρακτήων περιοχών. Ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη θάλασσα να απορροφήσει το διοξείδιο του άνθρακος όπως και τα τροπικά δάση. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, γιατί οι θάλασσες καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ποιες είναι οι δυνατότητες επιβίωσης για τους ωκεανούς, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις όλων αυτών. Δυστυχώς ο κύριος Μπρέχλεν δεν είναι παρόν, θα ήθελα να το ρωτήσω τι θα έπρεπε να κάνουμε για την προστασία της θάλασσας και τι θα έπρεπε να κάνουμε σε επίπεδο θαλάσσιας χωροταξίας. Ξέρω ότι η Γερμανία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο το οποίο έχει σαν στόχο να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με τις περιοχές του Natura 2000. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πώς θα μπορέσει να γίνει η χωροταξία στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Μπρέκλιν, ο οποίος είπε ότι δεν θέλει να υπάρξει ευκαμψία στην αρχή της ε, ε, σχετικής σταθερότητας. Βέβαια στη Γερμανία τους περισσεύουν οι υποστοστώσεις αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να του πω ότι εδώ θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην αλληλεία το ίδιο το οποίο ισχύει και για το, την αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή σεβασμός στους κανόνες της ενίας αγοράς. Λοιπόν, η επιμονή του στην ε, σχετική σταθερότητα σε μια χώρα όπου δεν εξαντλούνται οι ποσοστώσεις μου φαίνεται κάπως υπερβολική. Ούτως ή άλλως πάντως θα πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στους διάφορους ομιλητές. Πρώτα στον κύριο Σαφάντερ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκινώ με το θέμα των απορρίψεων. Σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρίαση και ήδη σήμερα γίνονται παράλληλα με τη σημερινή συνεδρίαση πολλές διαβουλεύσεις με τους αλληλείς. Εγώ δεν είμαι αλληλείας. Αλλά μπορώ να σας πω για τη μεταποιητική βιομηχανία. Θέσατε αυτό το ερώτημα των απορρίψεων, κυρία Βουλευτή. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Είναι ένα ταμπού, είναι ένα κοινό Το θέμα των απορρίψεων πολλές φορές το παρασιωπούμε. Τι να κάνουμε. Δεν έχει κανεί συμφέρον να το αναφέρετε το θέμα αυτό. Εμένα μου είπανε ότι σε κάποια περίπτωση απερίφθησαν 300 τόνοι στη θάλασσα. Φτάνουν τεράστιε ποσότητε, λοιπόν συνολικά οι απορρίψει. Πώ μπορούμε να λύσουμε τώρα το πρόβλημα αυτό. Καταρχήν θα μπορούσαμε να συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία για τους τόνους. Παραδείγματο χάρη πολλές φορές αλλιεύονται 30 τόνοι ενό θαλασσίου είδου και υπάρχει απόρριψη 10 τόνων βακαλάου. Πολλέ φορέ λοιπόν χάνεται ο βακαλάος αυτός και βέβαια μετακινούνται τα ψάρια αυτά οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πάντα την ίδια σύνθεση των αλλιευμάτων. Όλα αυτά οδηγούν σε μια μεγάλη σπατάλη πόρων και χρημάτων. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό για τα πλοία τα οποία αλλιεύουν στη Βαλτική και που αλλιεύουν μόνο ένα είδος δεν έχουν καμία δυνατότητα να είναι οικονομικά βιώσιμα. Ετέθη επίσης και το θέμα της περιφερικοποίησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση δεν έχω καμία αμφιβολία και εδώ ίσως θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια διαχείριση της περιφερικοποίησης η οποία να φτάνει μέχρι στους αλείς <clears throat> και μέχρι τη μεταποιητική βιομηχανία. Αυτά μπορούν να γίνουν μονάχα αν λαμβάνονται αποφάσεις εκ των κάτω προς τα άνω, εάν εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της μεταπληκτικής βιομηχανίας οι αλείς γιατί πολλές φορές γίνεται ουσιαστικά ένας Ολυμπιακός αγώνα για τα ψάρια. Είδαμε τι έγινε στις ΗΠΑ, Εκεί δεν υπήρχε μια σταθερή πολιτική και κάθε φορά αλλάζαν οι κανόνες. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια τεράστια κατασπατάληση φυσικών πόρων. Άλλες φορές υπάρχει και μείωση των τιμών των ηχθείων που οδηγούν σε δραματικές καταστάσεις για τους ε, αλείς ο στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι να εξετάσουμε το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο τους ε, ίδιους τους αλείς. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις λύσεις του 16ου, 17ου αιώνα όταν πήγαινε κανείς και αγόραζε στις ηχθειοσκάλες το ψάρι και δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός. Νομίζω τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση και θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και τη μεταποίηση. Για τα αλλιεύματα, εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με τους αλλείς. Αναφέρθηκε το θέμα του γάβρου, παραδείγματος χάρη, και, της, ε, και του ξηφία. Και στον τομέα αυτό υπάρχουν σημαντικές απορρίψεις. Αλλά για τη Βαλτική το κύριο αλλιευόμενο είδος είναι ο γάδος, που υπάρχει η δυνατότητα μονάχα να αλλιεύει κανείς ένα μήνα κάθε δύο, παραδείγματος χάρη οι αλλοί το έχουν δεχτεί και θα έπρεπε όμως να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν απαραίτητο να γίνει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ερώτηση της κυρίας Σάντσες Πρεσέδου πώς μπορούμε, του κυρίου συγγνώμη σαν σας πρισέδω, πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αύξησης των τιμών του καυσίμου, να σας πω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε εμεί καμία επιρροή στις ε, αλλαγές των τιμών. Και μάλιστα η επίπτωση είναι διπλώς αρνητική για μας, διότι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για παράδειγμα στις ε, ε, περιοχές ε, των ακτών για να αλλιεύσουν, αυτό που κάνουν είναι να περιμένουν να μειωθούν ε, περισσότερο οι τιμές και έτσι πλήττεται διπλά ο αλλιέας θα πρέπει να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για να, και να ε, λειτουργήσουμε συλλογικά για να μπορέσουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι είναι αλήθεια ότι ιστορικώς δεν υπάρχει τέτοια συνήθεια να αναλαμβάνουμε εμείς το ρόλο της, ε, τον εμπορικό Πρόκειται για οικογενειακέ επιχειρήσει, όπου συνήθω η γυναίκα είναι αυτή που αναλαμβάνει το εμπόριο. Αυτό που γινόταν παραδοσιακά ήταν ο άνδρας να ψαρεύει και η γυναίκα να πουλάει τα προϊόντα που Εμείς αυτό που μπορούμε να έχουμε είναι να έχουμε καλά προϊόντα στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να επιβραβεύονται και οι πρωτοβουλίες που πάνε, ε, προχωρούν υπέρ της βιωσιμότητας, τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε τις ε, αλλευτικές δυνατότητες, να προάγουμε και γραμμές χρηματοδότησης ε, για να βοηθήσουμε όλους όσους ασχολούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για κοινότητες αλλιευτικές οι οποίες προσπαθούν να βοηθήσουν στην ανάκτηση των πόρων και που στο κάτω-κάτω της γραφάς βρίσκονται σε αντίστοιχες συνθήκες με άλλες περιοχές οι οποίες δεν αναλαμβάνουν αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευχαριστώ. Πριν περάσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Μοντέιρα. Το ερώτημα λοιπόν ήταν η αλία πολλαπλών ειδών. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την έννοια της αηφορίας και την έννοια της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης όταν μιλάμε για αλληλεία πολλαπλών ειδών και όπου όλα αυτά τα είδη εγγράφονται σε ένα και το ίδιο οικοσύστημα. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν λειτουργικά να εφαρμόσουμε αυτή την έννοια στο μέλλον του MSY, την εφαρμογή της αρχής της ε, της βιώσιμης απόδοσης όταν μιλάμε για ένα συνολικό οικοσύστημα. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η εφαρμογή, αλλά αυτό μας φέρνει μπροστά σε ένα νέο δίλημα. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό κατά είδο ή πρέπει να το κάνουμε στα πλαίσια ενό οικοσυστήματο. Είναι διαφορετικό λοιπόν τα θέματα παραγωγικά τη θνησιμότητα των ειδών είναι διαφορετικά όταν μιλάμε για μεμονωμένα είδη και όταν μιλάμε για ένα συνολικό οικοσύστημα. Αυτό μα οδηγεί λοιπόν σε μια διαφορετική προσέγγιση. Ελπίζω ότι έχω απαντήσει επόμενο στο ερώτημά σα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Θέλετε να πείτε κάτι. Μετά από τις επιθέσεις των οποίων τύχατε από ορισμένου ομιλητές. Μερικοί ήταν καλοί, μερικοί κακοί και μετά <laughs> από την συνήκη της Λισαβόνας είπαν ότι εναποθένουν τις ελπίδες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σας συγχαίρω για αυτό το άριστο πάνελ ομιλητών με ποικιλία. Άλλοι υποστήριξαν την Κομισιόν, άλλοι την επέκριναν. Εμείς ακούσαμε και τα καλά νέα και τα κακά νέα. Αφήνουμε στην άκρη αυτά τα κάπως υπερβολικά, γιατί ό,τι είναι υπερβολικό είναι και ασήμαντο, όπως ξέρετε. Λογικό είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ να είναι επίδικη. Ωστόσο αυτή η ακρόαση οργανώθηκε πάρα πολύ καλά Είδαμε πρόσωπα που συνήθως βλέπουμε συχνά είτε στα ΡΑΚ, ή στην ΑΚΦΑ ή σε εξειδικευμένες συνεδριάσεις. Ο κύριος Δεμπένο, ο διευθυντής μου, το πρωί μου είπε ότι είναι πάρα πολύ στις συναντήσεις αυτές Και ο διευθυντής μου το πρωί ανάφερε τον προβληματισμό, μικρή αλληλεία, επιδοτήσεις, πρόσβαση, η προσπάθεια ως προς τις ποσοστώσεις. Φυσικά ξέρετε ότι η Κομισιόν πάντα ακούει. Η διαβούλευση θα κλείσει στο τέλος του μήνα. Θα καταλήξουμε σε πορίσματα το Μάρτιο, όταν θα έχει γίνει η πλήρης ανάλυση. Για να αντιδράσω όμως εν θερμό σε μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Η Κομισιόν σημείωσε το ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπουμε προκειμένου να μειωθεί το υπερβάλλον δυναμικών η πρόσβαση σε δικαιώματα μεταβιβάσεων μπορεί να βοηθήσουν με ξέρεση τη δανεία αλλά ταυτόχρονα και η ανάγκη προστασία σωσμένων μορφών αλληλείας ως προς κίνδυνο συγκέντρωσης ιδιαίτερα όσον αφορά τη μικρή αλληλεία. Δηλαδή εμείς συσχετίζουμε αυτά τα τρία στοιχεία της ΚΑΛΠ, υπερβάλλον δυναμικό, πρόσβαση στα δικαιώματα, ενδεχομένως μεταβιβάσιμα, αν και βέβαια θα πρέπει να ορίσουμε κάποια στιγμή σε τι επίπεδο γίνεται αυτή η μετάβαση. Είναι μια μετάβαση που γίνεται μέσα σε ένα κράτος μέλος ή μεταξύ κρατών, γιατί αλλάζει εντελώ το θέμα ανάλογα με το που, ξεκινάμε. Και τρίτον, τι επίπτωση θα έχει αυτή η μεταφορά στον κίνδυνο συγκέντρωσης δικαιωμάτων, άρα στη βιωσιμότητα της μικρής αλίας, η οποία σημειωθείται ότι πρέπει να προστατεύεται. Παρατήρηση για την ανανέωση του στόλου. Εδώ κανένας δεν έχει αντίρρηση. Μπορεί ο κάθε να ανανεώσει το σκάφος του, αλλά δεν αναφέρεται η ανανέωση του στόλου με δημόσιες ενισχύσεις. Όλοι εδώ μιλάνε για ανακαίνιση του στόλου, αλλά έχουν κατά δημόσιες ενισχύσεις. Η Κομισιόν όμως φυλάει ως κόριο οφθαλμού, είναι η μεταρρύθμιση του 2002, απαγόρευση ενισχύσεων για την ανανέωση, ανακαίνιση του στόλου. Εξεχρονισμός, ναι. Ενίσχυση για τα αλλιευτικά εργαλεία, ναι. Αλλά η ενίσχυση για ανανέωση των σκαφών, όχι. Το απαγορεύει η μεταρρύθμιση του 2002. Και η Κομισιόν δεν σκοπεύει να αναθεωρήσει αυτή τη στάση της. Αντίθετα, δεχόμαστε το ότι το υπερβάλλον δυναμικό να μην είναι ένα γενικό φαινόμενο, όπως είπαμε το 92 και όπως λέει και η έκθεση Γκέλλαν, μετά Λάσεν, ότι έχουμε υπερβάλλον δυναμικό 40%. Σήμερα η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Υπάρχουν ορισμένα επίπεδα που είναι σε ισορροπία, σε άλλα επίπεδα έχουμε μεγάλο υπερβάλλον δυναμικό. Πολύ μεγάλο στην Αγία Φερρυπίν του Μπακαλιάρου στη Βαλτική από τον Πολεμικό του Γάδου, συγγνώμη στη Βαλτική όπως μας ανάφεραν οι Πολωνία εδώ έχουμε ένα υπερβάλλον δυναμικό πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει κάπως να ρυθμιστεί η αποκέντρωση θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον διαδικαστικό επίπεδο, στρώμα συμφωνούμε κοιτάμε να δούμε τι γίνεται ως προς την δυνατότητα η εξουσία, η μάλλον στοιχεία εξουσίας γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τη συνθήκη που ορίζει ότι οι εξουσίες είναι στα χέρια των τριών θεσμικών οργάνων άρα ό,τι κάνουμε δεν θα πρέπει να διαταράσει το πνεύμα της συνθήκης περιφερειοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Να μην ισχύει για τους μακρινούς στόλους λόγω της φύσης της δράσης τους και τι σχέση έχει αυτή τους η δραστηριότητα με άλλους φορείς εκτός της Ένωσης. Το σημειώσαμε και αυτό. Είναι σημαντικό όσον αφορά την περιφερειοποίηση στη διαμόρφωση κανόνων ή στην εφαρμογή τους ποσόστηση, ε, πέρασμα μάλλον από προσπάθειες σε ποσόστοση για μεικτές δραστηριότητες. Έχουμε επίγνωση του προβλήματος, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα με τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις και πρέπει να βρούμε λύσεις. Ο κύριος Άμστρον πριν αναφέρθηκε σε ποσοστώσεις πολλών ειδών. Ενδεχομένως σε βάρος του πιο ευαίσθητου είδους. Πάντως, η προσφυγή στην έννοια MSWA πόλη είδους θα μας οδηγούσε σε ένα επίπεδο προσπάθειας που θα εκμεταλλευόταν σωστά ορισμένα θέματα υπερεκμεταλλευόμενοι, υποεκμεταλλευόμενοι συναφή ήδη και αποθέματα με τα ίδια αλλιευτικά εργαλεία. Οι ορισμοί, δύσκολο κεφάλαιο, καλύτερα θα είναι να μας βοηθήσουν οι κυβερνήσεις στους ορισμούς. Τι ισχύει για τις δικές τους παράκτιες ζώνες. Συμφωνούμε. Στόχος είναι ο στόλος μας να είναι αποδοτικός οικονομικά και ανταγωνιστικός. Αυτό όμω δεν συμφωνεί με ένα σύστημα ενισχύσεων που ζητάνε ορισμένοι, ζητάνε να διαιωνιστεί. Συμφωνώ με την κυρία Φράγα ότι αυτό που ζούμε είναι, η, αυτό που θέλουμε η οικονομική βιωσιμότητα των στόλων και όχι το να διαιωνιστούν οι κρατικέ ενισχύσει. Αυτό το λέει η πράσινη βίβλος. Αυτό που έθεσε ο κύριος Μπρελίνγκ ότι δηλαδή ορισμένοι αλληλείς και ο κύριος Στόβαν Στίβενσον το ανάφερε επίσης ότι υπόκεινται σε υποχρεώσεις στην περίπτωση του σχεδίου ανάκαμψης του γάδου χωρίς να έχουν ψερεύσει ούτε ένα γάδο. Παραξενεύουμε γι' αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Θα σας απαντήσω αργότερα, δεν θεωρώ δυνατό δραστηριότητα αλίας για ένα αλφα άλλο ψάρι ας πούμε θα μπορούσαν να συνεπάγονται υποχρεώσεις όρων που ορίζονται από το σχέδιο ανάκαμψης του γάδου. Στην κυρία Πάτρο Νέβε, στην εισηγήτριά σας, η Κομισιόν, είμαστε στη διάθεσή σας στην περαιτέρω επεξεργασία της έκθεσής σας για την μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ μου μένει μονάχα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν συμβάλει σε αυτή την πρώτη ακρόαση για το μέλλον της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Στο μέλλον του χρόνου συγκεκριμένα θα έχουμε πιο λεπτομερείς και λεπτομεριακές και πιο εστιασμένες ε, ακροάσεις. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ήδη από σήμερα μπορούν να αντιληθούν κάποια συμπεράσματα και κοινά στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν στις εργασίες της και νομίζω ότι υπάρχει λιγότερη απόκληση απόψεων από ό,τι θεωρούσαμε όλοι μας. Νομίζω ότι για τα βασικά στοιχεία μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια σαφή συμπεράσματα που θα λάβουμε υπόψη στην εκπόνηση της έκθεσης της κυρίας Πατράου. Αυτά λοιπόν θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα ανοιχτό φόρουμ για να παρακολουθήσει τα θέματα αυτά, να είναι πάντα στη διάθεσή σα για συζητήσεις και προφανώς με τους εκπροσώπους που ήταν παρόντες σήμερα θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας για μια καλύτερη πολιτική αλία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους και έχει τελειώσει η σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και απλώς πρέπει να ακολουθήσω τα σημεία της σημερινής διάταξης ενώ φεύγουν οι καλεσμένοι μας στο σημείο 16 στα διάφορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να θίξετε. Εάν όχι, έχει κλείσει και το σημείο αυτό και το σημείο 17 ανακοινώσεις της Προέδρου για αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από τους συντονιστές Νομίζω ότι ξέρετε ποια είναι τα συμπεράσματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και η επόμενη συνεδρία μας είναι 27-28 Ιανουαρίου το 2010. Μέχρι τότε, εάν δεν σας δω, σας εύχομαι καλές διακοπές και καλό νέο, καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ και τους διερμήνες και τέλος της συνεδρίασης.